Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με τη συνεδρίασή μας. Το σημείο 10 είναι το πρώτο στην ημερήσια διάταξη με την παρουσίαση του έργου ΕΣΠΟΝ Ευρωπαϊκό Δίκτυο Παρατήρησης Χωροταξιακού Σχεδιασμού με τον κύριο Μέλμπι και τον κύριο Σλάχτα, εμπειρογνώμονα για την Πολωνία. Και αυτό είναι και το ζήτημα ότι έχω αυτό το φοβερό MCRIT, αυτό το ακρονίμιο ε, στις σημειώσεις μου. Ε, ε φαντάζομαι ότι ο κύριος Σούλη θα μου εξηγήσει τι σημαίνει πρώτα απ' όλα. Αλλά μάλλον πρώτος θα λάβει το λόγο ο Πίτερ. Σε παρακαλώ, θα λάβεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ και την ε, Επιτροπή σας που μας επέτρεψε να έρθουμε να σας παρουσιάσουμε μια πολύ σημαντική και ιδιαίτερη εργασία, ένα έργο σημαντικό πιστεύω και για το Κοινοβούλιο και ειδικότερα την Επιτροπή σας. Ίσως ε, θα ήταν ο σκόπος να σας εξηγήσω πρώτα απ' όλα γιατί αποφάσισαν όλες αυτές οι χώρες, 32 τον αριθμό, να ε, ιδρύσουν αυτό το σχέδιο, να ξεκινήσω αυτό το σχέδιο, ε, λόγω καταρχάς των ζωφερών προοπτικών με την οικονομική αλλαγή, με την επίδραση του κλίματος, με την παγκοσμιοποίηση, με τις δημογραφικές πιέσεις, τη γύρενση του πληθυσμού στην Ευρώπη και τις μεταναστευτικές ροές διαφόρων τύπων, ε, με τις ενεργειακές προκλήσεις, και βέβαια με δεδομένη την επέκταση της ευρωπαϊκής επικράτειας. Βήμα το βήμα, που σημαίνει ότι πρέπει να δίνουμε πλέον απόκριση και σε εντυνόμενες αποκλίσεις μεταξύ των, του επίπεδου που γνωρίζουν διάφορες περιφέρειες στην Ευρώπη. Όλα αυτά λοιπόν ως υπόβαθρο της απόφασης και της επιλογής της θεματολογίας για το έσπρον. έσπον. Και έτσι αποφασίσαμε να αναπτύξουμε αυτό το project, το έργο που ονομάζεται σενάρια και οράματα και όραμα για το 2050 με βάση την πεποίθηση ότι μπορεί οι εδαφικές, οι εδαφικές δομές να είναι πολύ διαφορετικές και αποκομμένες, μπορεί κανείς να δείξει με ευφύ τρόπο και φάνταστο το δρόμο για το μέλλον και να προτείνει λύσεις που θα φέρουν αποτελέσματα στις περιφέρειες, αποτελέσματα τα οποία θα καρποθούν και οι προσεχείς γενιές. Αυτή είναι η βασική μας ιδέα. Για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του έργου έχουμε να κάνουμε με ένα ε, συνεκτικό πλαίσιο πολιτικών, ε, με καλύτερη αντίληψη του τι θέλουμε για το μέλλον. Δηλαδή, πρόκειται για μια προσπάθεια για δημιουργικότητα, για οραματικότητα, για χάραξη οραμάτων με στρατηγικό χαρακτήρα, οραμάτων που μπορούν να αποτελέσουν ένα πλαίσιο αναφοράς. Η light build όπως λένε στα γερμανικά, του διαλόγου για την πολιτική, για τη λήψη αποφάσεων από τους πολιτικούς και όχι μόνο στο τομέα της συνοχής θα έλεγα, αλλά και σε κάθε τομέα πολιτικής που μπορεί να έχει ε, αντίκτυπο στις περιφέρειες. Και άρα βλέπουμε μια προσπάθεια η οποία θα μπορούσε με τα οράματά της και έμεσα ακόμη να επηρεάσει αποφάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την οργάνωση των περιφερειών. Αυτά λοιπόν αποφάσισε η Επιτροπή Επιτήρησης. Έχουμε να κάνουμε με πέντε βήματα. Καταρχάς αναπτύ... αναλύουμε την κατάσταση, ως προς περιφέρειες Ευρώπης. Μετά έχουμε μία βάση σαν σενάριο με ορίζοντα το 2050, ποσοτική μάλλον ε, απόπειρα σχεδιασμού. Η ομάδα δε που έχει επιληφθεί του έργου και θα σας παρουσιάσω σε λίγο αναλαμβάνει και το τρίτο βήμα που είναι ο σχεδιασμός των περιφερειακών αυτών σεναρίων, τριών τον αριθμό και επί τη βάση αυτών οικοδομούμε ένα όραμα περιφερειακό για την Ευρώπη χωρικού σχεδιασμού το οποίο μπορεί να αξιοποιήσει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή σας και το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια συνένεση, αποδοχή από διαφόρους εμπλεκομένους στον τομέα αυτών φορείς. Είναι μια απόπειρα να δούμε σε ποιο βαθμό μπορούμε να ανταποκριθούμε στις ε, ε, προσδοκίες της ε, Επιτροπής Επιτήρησης. Και ακολουθεί το πέμπτο βήμα που αντίστροφα πια κοιτάμε έχοντας ορίσει τους στόχους πώς θα φτάσουμε σε αυτούς. Πώς μπορούμε δηλαδή να μετακινήσουμε το ευρωπαϊκό, την ευρωπαϊκή επικράτεια, την, ε, το χωρικό σχεδιασμό, ώστε να προσαρμοστεί στο όραμα. Είναι ένα αντίστροφο μοντέλο δηλαδή. Πάντως θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι είναι συμμετοχικής διαδικασίας Ένα έργο το οποίο αφού έχει γίνει αυτή η συζήτηση και η ανάπτυξη των διαφορών σεναρίων έχει οριμάσει, έχει προχωρήσει και μπορούμε να έχουμε ομάδες εργασίας, να προχωρήσουμε ακόμη και σε μια μεγάλη διάσκεψη στις αρχές της ε, Άνοιξης του 2014. Την οποία θα θέλαμε να προσκαλέσουμε και μέλη της Επιτροπής σας να συμμετάσχουν και γενικότερα στο διάλογο αυτό. Θα σταματήσω εδώ. Και αν μου επιτρέπετε θα δώσω το λόγο στους δύο από τους εταίρους του έργου αυτού της ε, ΕΣΠΟΝ. Δεν έχουν λάβει εργολαβικά εκ των 11 εταίρων ε, ανά την Ευρώπη, οι δύο είναι εδώ παρόντες, με πρώτο τον επικεφαλής, κύριο Ούλιτ από την Κρήτ και δεν θα σας πω τι σημαίνει. Και βέβαια μετά ο κύριος ε, Γιάτζεξ Λάξα θα αναλάβει να παρουσιάσει το υπόλοιπο κομμάτι. Σας σταματώ εδώ λοιπόν και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πέτρο. Ο κύριος Ούλιτ όπως μας είπατε θα εξηγήσει τη δραστηριότητα της εταιρείας του που ασχολείται με θέματα υποδομών. Πρώτα εκείνος λοιπόν και μετά ο καθηγητής Ζάχτα. Έτσι δεν το είπαμε με αυτή τη σειρά. Ωραία. Ο Ανδρέας Γούλιτ. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα. ναι, Αντρέα Σούλιτ λέγομαι και εργάζομαι στο ΜΚΡΙΤ που σημαίνει κριτήρια ή πολλαπλά κριτήρια. Κρίτ δηλαδή. και δράζεται στη Βαρκελόνη. Υγούμαστε 11 ερευνητικών ιδρυμάτων και πανεπιστημίων σε ολόκληρη την Ευρώπη για αυτό το έργο. Στην παρουσίασή μας αυτή θα τονίσουμε ιδιαίτερα τρία θέματα. Πρώτον, η περιφερειακή χωροταξική δυναμική μέχρι το 2030, δεύτερον ανάλυση εναρίνου για την Ευρώπη μέχρι το 2050 και τέλος η πιθανή νέα γενιά πολιτικής συνοχής. Αυτό είναι το πιο δύσκολο. Χαίρομαι που είναι εδώ και ο καθηγητής Ζάχτα που θα σας μιλήσει για τα συμπεράσματα και τις ιδέες μας. <clears throat> Ας αρχίσω λοιπόν με το πρώτο. Για να προβλέψουμε το μέλλον χρησιμοποιούμε ορισμένα μοντέλα μέχρι το 2050 για πολλαπλούς τομείς. Ο πίνακας που βλέπετε εδώ είναι το κύριο συμπέρασμα της μελέτης μας. This, uh, Αυτή η πρόβλεψη έγινε με βάση τις συνθήκες που ισχύουν σήμερα χωρίς να προβλέπονται αλλαγές στην πολιτική της κυρίαρχης τάσης. Αν δεν αλλάξει λοιπόν τίποτα στην εξέλιξη των πραγμάτων τότε έτσι θα είναι η Ευρώπη από περιφερειακής απόψεως. Βλέπετε ότι γενικά υπάρχει ένα ΑΕΠ 1,89% που προβλέπεται μέχρι το 30 είναι μέτρια ανάπτυξη, δεν θα την έλεγα χαμηλή, αλλά έχουμε και 45 περιφέρειες κάτω από 1% κατά μέσο όρο. Αυτές είναι οι κίτρινες και κόκκινες. Στα μπλε είναι οι περιφέρειες με χαμηλή ανάπτυξη και στο βαθύ Κιανούν είναι η ανάπτυξη 1,5 περίπου της 100 ΑΕΠ. Γενικότερα όμως το βασικό συμπέρασμα της πρόβλεψης αυτής βασίζεται σε δύο πράγματα. Ένα, πολλές νότιο-ευρωπαϊκές περιφέρειες δεν θα καταφέρουν μέχρι το 30 να ξεπεράσουν την κρίση. Και γι' αυτό αναμένουμε πολύ άσχημες καταστάσεις εκεί. Η ανάκαμψη θα είναι πολύ χαμηλή. Σύμφωνα με την πρόβλεψή μας θα είναι χαμηλότερη από εκείνη που προβλέπουν άλλες μελέτες εθνικές. Δεύτερο επίσης πολύ ανησυχητικό συμπέρασμα είναι ότι οι, Ανατολ... οι περιφέρειες της Ανατολικής Ευρώπης δεν αναπτύσσονται όπως οι δυτικές δηλαδή. Δεν έχει γεφυρωθεί το χάσμα. Αυτά είναι τα δύο αρνητικά συμπεράσματα από αυτή την πρόβλεψη. Υποθέτοντας βέβαια ότι δεν θα υπάρξει αλλαγή πολιτικής και θα συνεχίσουν τα πράγματα ως έχουν. Δεν είναι πιθανό να είναι τα πράγματα όντως έτσι το 2030, αλλά τα επόμενα χρόνια ναι. Τώρα αν συγκρίνουμε την πρόβλεψη αυτή με τις προβλέψεις του Δουνουτού μέχρι το 2017, όχι 30 όπως εμείς, βλέπουμε ότι η πρόβλεψη εκείνη δείχνει ακόμα χειρότερα συμπεράσματα για τις μεσογειακές περιφέρειες, αλλά πιο θετικά για τις ανατολικοευρωπαϊκές χώρες. Στη δική μας ανάλυση, συγκρίνοντας και τις δύο προβλέψεις, βλέπουμε ότι είναι πιο συμβατές μεταξύ τους από ό,τι φαίνεται εκ πρώτης όψεως. Δηλαδή, στην κόκκινη γραφική παράσταση βλέπετε τι συμβαίνει στις νότιες περιφέρειες και στην γαλάζια στις ανατολικοευρωπαϊκές. Βλέπετε ότι και οι δύο προβλέψεις από το Δουνουτού μέχρι το 17 και η δική μας μέχρι το 2030 μπορούν να συνδυαστούν. Βέβαια επειδή εμείς βασιζόμαστε σε περιφερειακό επίπεδο ίσως οι προβλέψεις μας είναι πιο λεπτομερείς και γι' αυτό είναι πιο απεσιόδοξες. Τώρα η δημογραφική εξέλιξη μέχρι το 2030. Επιβεβαιώνονται εδώ και άλλες προβλέψεις, δηλαδή στο κόκκινο, στις κόκκινες περιφέρειες μειώνεται ο πληθυσμός. Αν και παραμένει περίπου σταθερός ο ευρωπαϊκός πληθυσμός με πολύ λίγη αύξηση, υπάρχουν σημαντικές περιφερειακές διαφορές. Η Γερμανία ιδίως χάνει πληθυσμό και άρα μάλλον θα υπάρξει μεταναστευτική ροή προς τα εκεί και την Ανατολική Ευρώπη, γενικότερα ιδιαίτερα όμως στην Ευρώπη, στη Γερμανία. Τώρα η γύρανση του πληθυσμού είναι κοινό, κοινή τάση για ολόκληρη την Ευρώπη. Δεν θα έλεγα όμως ότι είναι προβληματικό αυτό γιατί η μείωση του πληθυσμού είναι πρόβλημα για τις περιφέρειες αλλά η γύρανση είναι διαφορετικό πράγμα και διαπαιτεί διαφορετική πολιτική κάθε αυτό δεν είναι πρόβλημα. Για να συνοψίσω λοιπόν όλες αυτές τις αναλύσεις. Βλέπουμε ότι θα ζήσουμε σε μια Ευρώπη με πολύ μεγάλες περιφερειακές ανισότητες. Εδώ σε αυτό το χάρτη βλέπουμε την εξέλιξη των προηγουμένων ετών. Στο μπλε περιφέρειες που αναπτύσσονται άνω του μέσου όρου, στα κόκκινα που αναπτύσσονται αλλά κάτω. Αυτό βέβαια είναι πλασματική εικόνα γιατί στο μέλλον αναμένουμε κάτι πολύ διαφορετικό. Αναμένουμε δηλαδή οι περιφέρειες με σταθερή και ισχυρή οικονομία να αναπτυχθούν κατά μέχρι και 2% ενώ εκείνες που έχουν λιγότερο αναπτυγμένη οικονομία να αναπτυχθούν λιγότερο. Η άλλη τάση που αναλύουμε είναι η διαφοροποιημένη παγκοσμιοποίηση. Δηλαδή με την κρίση βλέπουμε τις μετεγκαταστάσεις των ευρωπαϊκών εταιριών και εδώ είναι η συνδυασμένη εικόνα των επενδύσεων στην Ευρώπη. Βλέπουμε ισπανικές εταιρείες να επενδύουν στη Λατινική Αμερική, αγγλικές στις χώρες της κοινοπολιτείας, γερμανικές στην Ασία Υπάρχει λοιπόν αυξημένη διαφοροποίηση των εξωτερικών επενδύσεων των ευρωπαϊκών εταιριών και αν δούμε την εξέλιξη βλέπουμε ότι στη Γερμανία τώρα που είναι η πιο δυναμική περιφέρεια εξάγει πολύ στην Ευρώπη αν και δεν αυξάνονται οι εξαγωγές. Η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία είναι η Ισπανία η οποία επίσης αυξάνει τις εξαγωγές της εκτός Ευρώπης αλλά μειώνει τις εισαγωγές της από τις ευρωπαϊκές χώρες. Άρα όλο και περισσότερες δραστηριότητες ευρωπαϊκών εταιριών γίνονται εκτός Ευρώπης, μειώνονται εκτός Ευρώπης. Αυτό είναι διαφορετικό από ό,τι συνέβαινε τις τελευταίες δεκαετίες βλέπετε εδώ γενικότερες αλλαγές τα τελευταία 20 χρόνια που μάλλον θα ενδυναμωθούν στο μέλλον θαλάσσιες επικοινωνίες και ότι το εμπόριο μεταξύ βορείων λιμένων και ε, βορειοαμερικανικών πριν από 20 χρόνια ήταν κυρίαρχη συναλλαγή. Σήμερα όμως μόνο 5 εκατομμύρια τέους κυρίως από τη Βόρεια Αμερική προς την Ευρώπη. Αυτό δημιουργεί νέες προκλήσεις για τα κέντρα υπολογισμού γιατί ίσως να πρέπει να ξαναυπολογίσουμε από την αρχή, να επανεξισορροπήσουμε τα πράγματα. Ίσως πιο παραγωγικό θα ήταν λοιπόν για την Ευρώπη να υπάρξει αυτή η επανεξισορρόπηση όπως έγινε στις ΗΠΑ. Εδώ βλέπουμε τις διπυρωτικές αεροπορικές συνδέσεις. Υπάρχουν ευρωπαϊκά hub, το Παρίσι, το Σίπολ, το Χίθρο η Φραγκφούρτη. που κυριαρχούν στις αεροπορικές επικοινωνίες. Εδώ ο χάρτης δείχνει την χωροταξική πόλωση σε μερικά τέτοια κέντρα βασίζεται κυρίως στις γνωστές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες που έχουν μεγάλα αεροδρόμια αλλά και σε περιφέρειες κοντά στη Βαρκελόνη και τη Μασαλία που έχουν μεγάλα λιμάνια. Για να συνοψίσω λοιπόν αυτές τις περιφερειακές τάσεις θα έλεγα ότι μέτρια οικονομική ανάπτυξη, αύξηση των περιφερειακών ανισοτήτων, περισσότερες δουλειές με χαμηλότερους μισθούς. Δηλαδή, αν και η οικονομία είναι αδύνατη, ιδίως στις ανατολικές και νότιες χώρες, επειδή μειώνονται οι μισθοί, μπορούν να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις απασχόλησης. Περισσότερη κινητικότητα λοιπόν και μεταναστευτικές ροές από περιφέρειες προς το κέντρο γύρανση του πληθυσμού, διαφοροποιημένη παγκοσμιοποίηση και πόλωση σε ορισμένα αεροπορικά και λιμενικά κέντρα. Αυτά μπορέσαμε να μετρήσουμε. Το δεύτερο τμήμα τώρα. Σενάρια για το 2050. Αυτά είναι τα τρία σενάρια που έχουμε, στα οποία έχουμε καταλήξει. Το πρώτο το λέμε Promotion of Global Regions και δείχνει ορισμένες από τις τάσεις που ήδη αναφέραμε. Να ενισχυθούν δηλαδή τα κύρια αστικά κέντρα και ποιες είναι οι συνδέσεις μεταξύ τους. Αυτό το καθορίζει κυρίως η αγορά. Δεύτερον, εξισορρόπηση μέσω προώθησης μεγάλων περιφερειών και τρίτον σενάριο μεγαλύτερη αποκέντρωση του συστήματος. για μεγαλύτερη στήριξη της υπαίθρου. Αυτά είναι τα τρία ιδεώδη ακραία σενάρια που καθορίσαμε. Και μετά αναλύσαμε τα τρία αυτά σενάρια και τα συγκρίναμε σε διάφορες συνθήκες. Ακόμη και αν η οικονομία δεν λειτουργεί καλά, λόγω της τεχνολογικής προοδού και αύξησης της παραγωγικότητας θέλαμε να δούμε αν θα είναι υψηλότερο το κόστος της ενέργειας και των αντιμετώπιση των κλιματολογικών αλλαγών. Αυτή είναι η αριθμή. Το σημαντικό είναι να ξέρουμε ότι εμείς αναλύσαμε κυρίως το θέμα των διαρθρωτικών ταμείων και ταμείων συνοχής και βασιστήκαμε σε ίδια πολιτική. Ότι βασίζονται η χορήγηση των κονδυλίων από αυτά τα ταμεία κυρίως στις μεγάλες πόλεις ή στα άλλα σενάρια που αναφέραμε μεγαλύτερη προώθηση περιφερειακών και υπεθρίων περιοχών. Και από εδώ βγάζουμε δύο συμπεράσματα. Εδώ φαίνεται η συνοχή ως προς την μείωση των ανισοτήτων. Η αλλαγή της κατανομής των ταμείων οδηγεί σε διαφορετικά συμπεράσματα. Το γάμα 2 είναι το σενάριο που προβλέπει ταχύτερη μείωση των ανισοτήτων, ενώ το α3 λιγότερο ταχεία και λιγότερο ικανοποιητική εξέλιξη. Και μόνο η κατανομή λοιπόν των ταμείων τα αλλάζει όλα. Και αυτό είναι κατανοητό διότι αν έχουμε την ίδια πολιτική εδώ και 20 χρόνια είναι λογικό να έχει αυτά αποτελέσματα. Αν και το συνολικό ύψος των μαντιλίων παραμείνει το ίδιο και μόνο από την διαφορετική κατανομή μπορούμε να καταλήξουμε σε μεγάλες διαφορές. Ταυτόχρονα όμως βλέπουμε ότι και τα τρία σενάρια συνεχίζουν με την ίδια τάση. Η μείωση των ανισοτήτων, προσπάθεια που γίνεται εδώ και 20 χρόνια, θα συνεχίσει στο μέλλον μόνον εάν εφαρμοστούν πολύ πιο ριζοσπαστικά προγράμματα. Αυτά είναι τα δύο μηνύματα στα οποία καταλήξαμε. Και τελειώνω τώρα για να δώσω το λόγο στον καθηγητή. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ μόνο τρεις διαφάνειες έχω. Στην πρώτη διαφάνεια βλέπετε το όραμά μας το 2020 ως σημείο εκκίνησης στις 11 Οκτωβρίου στην Επιτροπή των Περιφερειών θα γίνει ένα σεμινάριο ΕΣΠΟΝ σε ό,τι αφορά τα οράματα αυτά. Θα σας καλούμε λοιπόν όλους σας. Ε. Ως τώρα από τις συζητήσει έχουν προκύψει τα παρακάτω σχόλια, παρακάτω ιδέες ε, σε σχέση με το πώς θέλουμε να αλλάξουμε το μέλλον μέχρι το 2050, όχι για μας, αλλά τα, για τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Καταρχάς, να ακολουθήσουμε μια πολυκεντρική προσέγγιση για να αξιοποιηθεί το δυναμικό όλων των περιφερειών. Κατά δεύτερον, να χρησιμοποιήσουμε τα πλανεκτήματα της ε, προηγμένης ενοποίησης. Να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν τα ευφυή δίκτυα, τις ευφυής περιοχές. Οι εταίροι μας θέλουν να υπάρξει ενοποίηση σε ό,τι αφορά την προσέγγιση για τις περιφέρειες και χρησιμοποιώντας ε, τα εκτίματα για τα ασφαλή αλλά και ευέλικτα σύνορα για την καλύτερη αξιοποίηση της δικτύωσης. Επίσης, να κοιτάξουμε τις περιοχές ως ε, περιοχές, τις περιφέρειες ως περιοχές με παγκόσμια ανταγωνιστικότητα. Με μια προσέγγιση βάσει την περιοχή. Περιφέρειες που θα έχουν τις δικές τους ε, δυνατότητες και το δικό τους δυναμικό. Ύστερα, προσβασιμότητα και συνδεσιμότητα. Όλες οι περιφέρειες να είναι εσωτερικά και εξωτερικά προσβάσιμες για τους επιχειρηματίες, τους τουρίστες, τους πολίτες, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και γενικά ε, για ασφαλείς επαφές το τοπίο, το πολιτισμικό τοπίο χρησιμοποιούνται σαν επιπλέον πλεονεκτήματα έχουν ένα πάρα πολύ, μια πολύ λέξη οι Γερμανοί, τη χωροταξία για τέτοια πράγματα. Και η οικολογική βιωσιμότητα, η κλιματολογική αλλαγή, η προσαρμογή βάσει των πράσινων τεχνολογιών και πολιτικών. Τρεις ε, διαφάνειες σας είπα θα χρησιμοποιήσω. Στη δεύτερη διαφάνεια βλέπετε την πρόεδρό με ένα σημαντικό συμπέρασμα σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα της ε, πολιτικής συνοχής στην Πολωνία. σε ό,τι αφορά και την αύξηση των διαφορών μεταξύ των περιφερειών της Ευρώπης, γιατί οι μακροοικονομικές διαφορές μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης ε, ήταν μεγάλες και αυτές οι περιοχές ήταν που επλήχθησαν πιο πολύ από όλες. Έχουμε πολλά θέματα σε ό,τι αφορά τη διαχείριση, σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές. Τρία ερωτήματα λοιπόν θέτουμε στην παρούσα φάση. Καταρχάς, οι περιφερειακές αυτές διαφορές πόσο θα αυξηθούν το 2018 μέχρι το 2030 σύμφωνα με τις ε, προβλέψεις μας θα συνεχίσουν να αυξάνονται οι διαφορές και μόνο μετά το 2030 θα μειωθούν. Ύστερα, τι επίπεδο οικονομικού περιθωρίου μπορούμε να προβλέψουμε μεταξύ των περιοχών, των περιφερειών με τις ίδιες νομικές, ε, νομικούς όρους. Οι διαφορές που υπάρχουν σήμερα είναι σε απαράδεκτο επίπεδο ουσιαστικά και θα αυξηθούν και όλα. Αυτό έχει ασφαλώς πολλές συνέπειες. Και τρίτη ερώτηση, πώς μπορούμε να περιορίσουμε τους πόρους της πολιτικής ε, την προγραμματική περίοδο μέχρι το 2020 έχουν προταθεί πολλές αλλαγές. Ελπίζω έτσι να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Ενδεχομένως να προσαρμόσουμε και τους τον κανονισμό να ακολουθήσουμε την περιφερειακή προσέγγιση να, να εφαρμοστεί η αστική πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η σχετική όρη της πολιτικής μέχρι το 2020. Αλλά οι εκχωρήσεις σε ό,τι αφορά την επόμενη πραγματική περίοδο, σε πολλές περιπτώσεις είναι σε αναλογία 2 προς 1. Επίσης, σε ό,τι αφορά τον γεωργικό κλάδο υπάρχουν θέματα. Και τώρα να περάσω στην τελευταία μου διαφάνεια. Τι γίνεται με τη νέα γενιά πολιτικών συνοχής μετά το 2020. Η πολιτική συνοχής που δεν αποδίδει συνοχή θα μπορούσε να αποτελέσει, αν θέλετε, στόχαστρο για τα βέλη της κριτικής. Καταρχάς, ε, ανάπτυξη του δυναμικού των τοπικών και περιφερειακών φορέων διοίκησης. Καλύτερη δικτύωση των φορέων αυτών. Και περιφερειακή προσέγγιση επενδύσεις ε, σε περιφερειακό επίπεδο να αντιμετωπίσουν τους πλειοτικά προγράμματα μόνο. Κατά δεύτερον, προώθηση της τοπικής ανάπτυξης, της ενδογενούς ανάπτυξης. Με τη χρήση των, του τοπικού δυναμικού. Δεν χρειαζόμαστε 55 Silicon Valley στην Ευρώπη, όχι. Θέλουμε η κάθε περιφέρεια να χρησιμοποιεί τα πλεονεκτήματά της, το δυναμικό που ήδη έχει. Κατά τρίτον, ευαισθησία σε ό,τι αφορά τους οικονομικούς κύκλους. Ευελιξία, προσαρμογή των πολιτικών, όπου αυτό είναι απαραίτητο. Όχι μόνο τους ε, ε, επιχειρησιακούς κύκλους, αλλά και τους κύκλους του Ταμείου Συνοχής κατά τέταρτον. Ε, μεγαλύτερη επικέντρωση σε ό,τι αφορά τα τοπικά και περιφερειακά συστήματα υποδομών. Κοιτάμε τι γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά σε πολλές περιοχές της Ευρώπης η εξωτερική αλλά και εσωτερική προσβασιμότητα θα πρέπει να υπάρχει και μάλιστα να έχει υψηλή ποιότητα. Πέμπτον, μέτρα και mm. μέσα αυστηρής χρήσης για τη γη σε ευαίσθητες περιοχές. Χρειαζόμαστε λοιπόν μεγάλης ποιότητας ε, σχεδιασμό και μέτρα για την ανανέωση έκτον. Ε, παραγωγικές επενδύσεις σε γειτονικές χώρες. Βλέπετε στο χάρτη ότι οι πιο ασθενείς, οι λιγότερο εύρωστες περιοχές είναι οι περιοχές ε, οι γειτονικές της ε, Ευρώπης. Άρα μπορούμε να δημιουργήσουμε και να εκμεταλλευτούμε την εγκύτητα για να ε, δημιουργήσουμε κέρδος για, αμφότερες πλευρές, και τις αμφότερες πλευρές των συνερών. Αυτά ήθελα να αναφέρω γιατί θέλουμε μέχρι τα μέσα του 2014 να ολοκληρώσουμε το project μας. Σας προσκαλούμε λοιπόν στις συζητήσεις μας. Ελπίζουμε και στο μέλλον να μπορέσουμε να έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για το πώς θα διαμορφωθεί καλύτερα η πολιτική συνοχή προκειμένου να έχει πραγματικά ως αποτέλεσμα τη συνοχή για την Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Και δεν θέλω να ξεκινήσω, μια και έχουμε λίγο χρόνο για ερωτήσεις και σχόλια, με τον κύριο Ολμπριχτ. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέρον το υλικό. Επίσης, τουλάχιστον να το διαβάσουν οι πολιτικοί και όσοι ασχολούνται με αυτές τις στρατηγικέ, να δουν ποια είναι η κατάσταση. Δύο ερωτήσεις. Η μία έχει πολιτικό, πολιτικό χαρακτήρα για τους εμπειρογνώμονές μας που δεν είναι υποχρεωμένοι να απαντήσουν με πολιτικούς όρους. Αλλά αν κοιτάξουμε το ΑΕΠ, κατά κεφαλήν ΑΕΠ, η ανάπτυξη είναι ορατή σε ορισμένες χώρες, αλλά μετά παρουσιάζει αντίστροφη Τι μπορεί να προσφέρει λοιπόν η περιφερειακή πολιτική με τέτοια περίπτωση. Δηλαδή, η πολιτική συνοχή τι μπορεί να προσφέρει. Ξέρετε ότι από τον περιορισμό των αποκλήσεων των διαφορών έχουμε περάσει στο ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και το καθεξής. Μήπως όμως τελικά έχουμε ξαναπέσει στη συζήτηση για τις πολιτικές που χρειάζονται ώστε να στηριχθούν αυτές οι χώρες και αυτές οι περιφέρειες που βρίσκονται σε πιο αδύναμη θέση. Και εδώ μιλάω για πολιτικές επιλογές, οι οποίες αναφέρονταν στο 2020. Η κατάσταση όμως αποδεικνύεται ότι εάν έτσι ε, ε, καταστάσεις όμως αποδεικνύεται ότι αν δεν βοηθήσουμε τους ε, πιο αδύναμους θα έχουμε περισσότερο κόστο και σε σχέση με τους πιο ε, Έγινε λοιπόν όλη αυτή η προσπάθεια για να ολοκληρώνω. Να πούμε ότι και να αποδείξουμε ότι η πολιτική τη συνοχή δεν είναι πολιτική συνοχή, αλλά επενδύσει για την ανταγωνιστικότητα. Και τώρα ξανακύλαμε πάλι στα ίδια. Τι χρειάζεστε λοιπόν. Και δεύτερον, Εδώ έχουμε να κάνουμε μια κατάσταση που έχει διαφορετική εικόνα μέσα στην Ευρωζώνη και άλλη στα 28 κράτη-μέλη τα ζητήματα με τα six-pack, με την αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα και το καθεξής σημαίνουν μια διαφορετική οικονομική κατάσταση για την Ευρωζώνη. Μήπως θα έπρεπε λοιπόν, αντί για τα σενάρια που μας παρουσιάσατε, να ε, σχηματίσετε ένα άλλο σενάριο το οποίο να δείχνει οράματα για τη δυναμική ε, πορεία της Ευρωζώνης και ούτω καθεξής. Τίποτα δεν έχει αλλάξει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, δεν ξέρω αν θέλει κανείς άλλο στο λόγο. Θέλω όμως εγώ να κάνω μια ερώτηση. Όταν ε, αναπτύσσω αυτά σενάρια για το μέλλον, για την Ευρωπαϊκή Επικράτεια, λέτε ότι θα υπάρχουν αυτό που ονομάζουμε περιφέρειες, ε, δάφη, συνολικά δηλαδή η θεώρηση των περιφερειών αυτών και το άνοιγμα στον κόσμο. Μιλάτε επίσης εν γέννη για τα αστικά κέντρα και μετά για τις περιφερειακές περιοχές, η περιοχές της Ευρώπης, της Υπέθρου. Αλλά δεν βλέπω να λέτε τίποτα για την αξιοποίηση διασυνδέσεων, συσχετισμών μεταξύ αυτών των διαφόρων ειδών περιφερειών που θέλετε να προαγάγετε. Δεν φαίνεται δηλαδή να κάνετε την επιλογή και την προσφορά ώστε να μπορέσουν να συνεργαστούν, να συνδεθούν μεταξύ τους, να έχουν μια κοινή πορεία. Θα κάνετε σχόλια σε αυτό. Αν δεν θέλει κανείς άλλο το λόγο, να ακούσω τα σχολεία σας. Ναι, ας ξεκινήσω με την τελευταία ερώτηση. Γιατί ναι, όντως βρίσκεται στο επίκεντρο των μελημάτων μας. Από τις ε, μελέτες που έχω κάνει στο παρελθόν και πριν από την κρίση. Περισσότερο, πρέπει να πω, είχαμε μέλημα αυτή την ε, διασύνδεση των ευρωπαϊκών οικονομιών βλέπουμε ότι όσο πιο στενή είναι η διασύνδεση, τόσο καλύτερα προχωράμε. Και για το παράδειγμα, το συγκεκριμένο, η Γερμανία ε, πουλούσε πολύ και η Ισπανία αγόραζε πολύ από τη Γερμανία, συμπεριλαμβανομένης και από της Γερμανίας. Άρα αυτή η ανάπτυξη ήταν ε, ωφέλιμη για τους πάντες. Μετά την κρίση όμως κατάσταση και η εικόνα είναι διαφορετική. Βλέπουμε δηλαδή πρώτα ότι ίσως δεν ήταν αηφόρο, δεν ήταν διατηρήσιμο στο μέλλον οικονομικά το φαινόμενο το οποίο είχε παρατηρηθεί. Ε, φάνηκε δηλαδή σαν να αγόραζαν περισσότερο από ό,τι θα μπορούσαν ε, να αντέξουν οικονομικά οι χώρες του Νότου. Και από την άλλη βλέπουμε ότι οι εθνικές οικονομίες, οι κοινωνικές οικονομίες ε, έχουν παγκοσμιοποιημένο χαρακτήρα πλέον. Επομένως μήπως πρέπει να ε, αναλογιστούμε ότι αυτές οι διασυνδέσεις που υφίστανται και υπάρχουν και τα συστήματα και οι νόμοι μεταφοράς και τα λοιπά ε, χρειάζονται διαφορετική θεώρηση γιατί υπάρχουν οι διασυνδέσεις. Επίσης για τις ε, γειτονικές στην Ευρώπη χώρες Νότια, ε, Βόρεια Αφρική, Ανατολική Γειτονία, πρώην χώρες ε, της Σοβιετικής Ένωσης. Ε, τις λοιπόν που έχει ο καθένας θα πρέπει να τις ε, λαμβάνουμε υπόψη πλέον πολύ περισσότερο από στο παρελθόν. Και για να καταλήξω, δεν φαίνεται να έχουν αυτές οι διασυνδέσεις τόσο στρατηγικό χαρακτήρα, διασυνδέσεις μεταξύ περιφερειών δηλαδή, όσο άλλου τύπου διασυνδέσεις. Και βεβαίω συμφωνούμε ότι υπάρχει κόστος από τον κατακερασματισμό στην Ευρωζώνη. Και ο κατακερματισμός για το χρέος που πληρώνει η Ευρώπη είναι τεράστιος για το χρέος που πληρώνει συνολικά η Ευρώπη σε σχέση με αυτό που πληρώνει η Κίνα, η Ιαπωνία και το καθεξής. Μιλούμε για στοιχεία κλειδιά που ενισχύουν την κρίση. Η Ευρωζώνη λοιπόν χρειάζεται ενίσχυση νέα, αλλά είναι δύσκολο να ισχυριστεί κανείς ότι η κατάσταση που έχουμε τώρα με τον κατακαιρματισμό της Ευρωζώνης είναι η καλύτερη λύση. Το να ενισχυθεί η Ευρωζώνη ασφαλώς θα αλλάξει τη γραμμή βάσης ε, και ελπίζω ότι θα την αλλάξει προς το καλύτερο. Το να υπάρξει καλύτερη ενοποίηση δηλαδή στην Ευρωζώνη, η αποφυγή του κινδύνου της, ε, του κατακαιρματισμού. Αν μου επιτρέπετε θα ήθελα και εγώ να συμπληρώσω κάτι σχετικό με την πρώτη ερώτηση του κ. Ολπριχτ. Όταν έλαβε ο ήλιος λαμπρός για την Ευρώπη, οι πιο αδύναμες περιφέρειες απομυζούσαν πλεονεκτήματα από την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και βλέπαμε ισχυρή την παρουσία και την, τον αντίκτυπο της πολιτικής συνοχής. Σαφές όμως καθίσταται μετά το 2008 ότι πιο αδύναμες περιοχές είναι πιο ευάλωτες στις αρνητικές μεγατάσεις έχουν δηλαδή χαμηλότερο δυναμικό απορρόφησης κλειδονισμών και ανέβρεσης των εξωτερικών πηγών ανάπτυξης. Και άρα θα πρέπει να αναλογιστούμε για άλλη μια φορά τι σημαίνει πολιτική συνοχής, και τι τμήματα θα έχει αυτή η πολιτική. Το πρώτο τμήμα της θα είναι ασφαλώς ε, προσανατολισμένο προς τη συνοχή, αλλά το δεύτερο περισσότερο προς την ανταγωνιστικότητα. Γιατί αν η κατάσταση όπως την έχουμε τώρα, η ανάπτυξη για την Ευρώπη, πολιτική, οικονομική, ε, χωροταξική, ε, περιβαλλοντική, θα είναι πολύ προβληματική και μπορεί να πλήξει και την, την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση κάποια στιγμή. Αυτή είναι η παρατήρησή μου. Σα ευχαριστούμε, Πίτερ. Ναι, για να απαντήσω λίγο τα ερωτήματά σας, να πω το εξή. Νομίζω ότι τα τρία σενάρια που μας ε, καταδείχθηκαν και στους χάρτες είναι ακραίες λύσεις, αν θέλετε. Ακραίες εναλλακτικές όταν κάνουμε τη συζήτηση για το τι θα μπορούσε να αποτελέσει το περιφερειακό όραμα για την Ευρώπη το 2050, στη διαδικασία θα πρέπει να βρούμε τη διασύνδεση και το σωστό μείγμα πολιτικών που μπορεί να εκφράσει ακριβώς τις σχέσεις αυτές. Μιλάμε λοιπόν για ακραίες εναλλακτικέ και αυτό το κάνουμε σκόπιμα, αλλά μέσω του διαλόγου θα πρέπει να τα συνενώσουμε όλα αυτά και να βρούμε το σωστό μείγμα. Ελπίζω έτσι να απαντάω στην ερώτησή σας. Συνάδελφοι, σας παρακαλώ, συνεδριάζουμε. Λίγη ησυχία. Ναι, συγγνώμη, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα, ίσως για όχι για τη δική μας Επιτροπή, αλλά για τη Μελλοντική Επιτροπή, γιατί η πολιτική συνοχής προγραμματίζεται εκ των προτέρων από πολύ πιο νωρί. Άρα για μα αυτά που θα συμβούν σε 15-20 χρόνια δεν είναι κάτι το αφηρημένο, ένα αφηρημένο πολιτικό όραμα. Όχι, πρόκειται για έναν παράγοντα που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μα εδώ και τώρα. Γι' αυτό λοιπόν μας ενδιαφέρει το τι γίνεται με το ΕΣΠΟΛ. Χτες είπατε ότι υπάρχει και αυτή η ιδέα για να ανταποκρινόμαστε σε αιτήματα των κρατών μελών σε σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά θεωρώ ότι όλα αυτά είναι πολύ απαραίτητα, γιατί πριν από κάποια χρόνια δουλεύαμε και προετοιμάζαμε τις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες το 2020. Θα πρέπει λοιπόν υπό αυτούς τους όρους να δουλεύουμε. Και αυτό που μου λείπει στην προσέγγιση σας είναι το να ψάξουμε ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες ανάπτυξης στις περιφέρειες ε, της Ευρώπης. Γιατί έως τώρα η δημογραφία ευνοούσε την ανάπτυξη, αλλά αυτό θα διστραφεί πλέον. Και η Ευρώπη έχει πολύ χαμηλό ποσοστό ανάπτυξης, όπως είπατε. Αυτό ασφαλώς και επηρεάζει πολλές πτυχές του δημόσιου βίου. Άρα, Προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθούμε και να δούμε ποιοι είναι οι παράγοντες ε, ανάπτυξης επί των οποίων θα πρέπει να επικεντρωθεί η πολιτική. Δεν ξέρω, ενεργειακή αποδοτικότητα ίσως. Νομίζω όμως ότι θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο να ακολουθήσετε και αυτή τη γραμμή στα σενάρια που καταρτίζετε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να πάρει το λόγο. Ο κύριος Δίξτρα. Ευχαριστώ. Σας κατευχαριστώ κυρία Χουμπνερ. Είμαι από τη Γενική Διεύθυνση Περίφ. Με συγχωρείτε συνάδελφοι, ε, μερικοί θέλουν να ακούσουν. Και ήθελα να κάνω μερικά σύντομα σχόλια για τις παρουσιάσεις. Πρώτον, είναι πολύ φιλόδοξη χρονική περίοδος που χρησιμοποίησαν. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς με από σήμερα να προβλέψει οτιδήποτε για το 2050. Άρα όλα αυτά είναι υποθετικά. Επίσης θέλω να τονίσω το εξής. Διαφωνώ βασικά με τις προβλέψεις που λένε ότι θα αυξηθούν οι περιφερειακές ανισότητες. Αν δούμε τις προβλέψεις του Δουνουτού δεν βλέπουμε τίποτα τέτοιο και γι' αυτό νομίζω ότι η πολιτική συνοχή συνεργάζεται με την αγορά. Είμαι πεπισμένος ότι η ενιαία αγορά θα συμβάλλει στη μείωση των ανισοτήτων στο μέλλον. Η πολιτική συνοχή είναι σημαντική αλλά δεν είναι ο κύριος παράγοντας. Τώρα για αυτά που είπε ο Γιάνν Όλμπρεχτ πρέπει να κάνουμε σαφή διαχωρισμό μεταξύ της χρηματοδότησης που θα κατανείμουμε στις περιφέρειες και της χρήσης τους. Εμείς τονίσαμε ότι τη σημασία του ανταγωνισμού αλλά ως εργαλείο η κατανομή της χρηματοδότησης στοχεύει στη σύγκληση και τη μείωση των ανισοτήτων. Βέβαια δεν αναμένουμε οι περιφέρειες να δαπανίσουν όλα αυτά τα κονδύλια μόνο για υποδομές αλλά και στη δημιουργία επιχειρησιακού κλίματος κλπ. Όλα αυτά είναι επίσης σημαντικά για την οικονομική ανάπτυξη. Τέλος, δεν νομίζω ότι πρέπει να στοχεύουμε στο ίδιο ΑΕΠ παντού, αλλά μια ισοδύναμη ποιότητα ζωής στις περιφέρειες. Μερικές θα είναι πάντοτε πιο ανταγωνιστικές από άλλες, αλλά αυτό μπορεί να μην είναι πρόβλημα αν έχουν υψηλή ποιότητα ζωής. Ευχαριστώ. Μα αυτό είπε και ο Γιάννη. Μεγαλύτερη κινητοποίηση της δυνατότητας ανάπτυξης για τη βελτίωση του ιδιωτικού επίπεδου των περιφερειών. Σύγκληση και δυνατότητα ανάπτυξης. Δεν ξέρω αν κανείς άλλος θέλει να απαντήσει, ίσως ο Πέτρος. Ναι, με τον Λουίς πάντοτε ενδιαφέρουσε συζητήσεις έχουμε, αλλά 90% των σχολείων σου τα δέχομαι. Ας μιλήσω όμως για το υπόλοιπο 10%. Το χειρότερο σενάριο που είπαμε, εσύ το βρίσκεις ε, ο μη ρεαλιστικό, αλλά αυτά τα υπολογίσαμε από την αρχή της κρίσης, δηλαδή συμπεριλαμβάνουμε και τις επιπτώσεις της. Και μετά συγκρίνουμε τα στοιχεία του Δουνουτού για το 17 με πρόβλεψη για το 30 που κάνουμε εμείς. Οι διαφορές μπορεί να είναι σημαντικές αλλά τελικά δεν καταλήγουν σε τόσο διαφορετικά συμπεράσματα τελικά. το αποτελ, τα αποτελέσματα της κρίσης στην Νότια και Ανατολική Ευρώπη ήταν πολύ αρνητικό. Υπάρχει στις περιφέρειες αυτές η μαύρη παράνομη οικονομία που μπορεί να φτάνει μέχρι και το 25% του ΑΕΠ σε πολλές από αυτές τις χώρες. Και στην Υπεθρογιατή Γεωργία η στην Ανατολική Ευρώπη, στη Γεωργία στην Ανατολική Ευρώπη και στις κατασκευές και τον τουρισμό στις νότιες. Στην επίσημη οικονομία δεν συμπεριλαμβάνονται όλα τα πραγματικά στοιχεία. Δεν βλέπουμε δηλαδή εξωτερικούς δείκτες ως προς τη σκληρότητα της κρίσης, αλλά ήταν σκληρία οι επιπτώσεις της. Και προσθέτω Κάτι που Επίσης είπε ο Λουίς και είναι σωστό ότι η οικονομία τα τελευταία 20 χρόνια ήταν πολύ θετική. Δηλαδή οι ανατολικοευρωπαϊκές και νοτιοευρωπαϊκές χώρες σήμερα είναι σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι τότε. Δηλαδή οι Ευρωπαϊκές χώρες θα αναπτυχθούν λίγο παραπάνω από το μέσο όρο αλλά και οι άλλες θα επιβιώσουν. Όλα αυτά είναι λεπτομέρειες αλλά μετά από όλα αυτά δεν θα έλεγα ότι η πρόβλεψή μας διαφωνεί με τις προβλέψεις τις υπόλοιπες τις εθνικές γιατί, και του Δουνουτού γιατί έχουμε άλλο χρονικό εύρος. Βέβαια κανείς δεν ξέρει το μέλλον και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να το φανταστούμε. Ευχαριστώ. Ο Πίτερ. Θέλω να ξαναευχαριστήσω την Επιτροπή που μας έδωσε το, την ευκαιρία να συζητήσουμε αυτό το έργο. Βέβαια όταν κοιτάζει κανείς τα στοιχεία, τα ποσοτικά τους αριθμούς, μπορεί να είναι θεωρητικά, εντάξει. Όσο πιο απομακρυνόμαστε από το παρόν τόσο πιο αβέβαια είναι. Αλλά το βασικό στοιχείο της μελέτης της πρόβλεψης είναι ότι κάνει και μία ποιοτική δημιουργική προσπάθεια να υπάρξει μια κοινή κατανόηση με τους πολιτικούς ως προς το τι μέλλον θέλουμε. Φυσικά χρειάζεται και μια ποσοτική βάση, αλλά το κύριο του επιχείρημα είναι ποιοτικό. Αυτό προσπαθούμε εμείς στο ΕΣΠΟΝ. για αυτή την κοινή κατανόηση του μέλλοντος. Και ελπίζουμε και τα μέλη της Επιτροπής σας στο μέλλον να μας βοηθήσουν για να δημιουργηθεί αυτού του είδους η κοινή κατανόηση για το 50. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Uh, Ευχαριστούμε ξανά το ΕΣΠΟΝ και ελπίζουμε πριν λήξει η θητεία μας να σας ξανακούσουμε Τώρα συνάδελφοι περνάμε στο επόμενο σημείο που είναι το 11 δηλαδή ψηφοφορίες. Ελέγξτε με τις μηχανές σας παρακαλώ και τις κάρτες σας. Αρχίζει μια ενδεικτική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ελέγχουμε παρακαλώ να βάλετε όλοι τις κάρτες σας. Ενδεικτική ψεύτικη ψηφοφορία. Όσοι δεν ξέρουν να πατήσουν οποιοδήποτε από τα τρία κουμπιά. Όποιο θέλουν, όποιο θέλουν. Μερικοί δεν θέλουν φαίνεται. Τέλος πάντων έλξη ψηφοφορία. Να μην παραπονεθούν όσοι δεν δοκίμασαν. Λοιπόν, έκθεση Βλάσακ. Ρόι Ευχαριστώ πολύ. Η έκθεση αυτή προετοιμάστηκε με μεγάλη φροντίδα και κατάλογο ψηφοφορία. Και ο κατάλογο ε, του ΕΛΚ. Να ζητήσω από τα μέλη να με ψηφίσουν και να ακολουθήσουν το, το πτυτικό πρόσημο στην ε, τροπολογία 10. Ε, υπάρχει ένα αρνητικό πρόσημο στη λίστα σε ό,τι αφορά τους συναδέλφους και τη δική μου άποψη. Ε, θεωρούμε ότι θα ήταν θετικό το πρόσωπο. Θα σας τα υποδείξω και την ώρα της πληροφορίας. πρόεδρο. Αυτά ήταν τα σχόλιά σα λοιπόν και μπορούμε να ψηφίσουμε μάλιστα. Ωραία. Ψηφίζουμε την τροπολογία 12 λοιπόν και την 8 των ε, προπολογισμού υπέρ. Επιτροπή προπολογισμών. Κατά. Αποχέ, απορρίπτεται. Και τώρα περνάμε στην τροπολογία 18. Ψηφίζουμε την 18 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τώρα 17 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην 7 της Επιτροπής Προπολογισμών υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Στην 9 υπέρ κατά απορρίπτεται 10 υπέρ κατά αποχές έγκρινεται 13 και η 9 της Επιτροπής Προεπιλογισμών ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 19 υπέρ Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τίτλος 1. Ε, budget 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Οι δύο της Επιτροπής Προλογισμών υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. λογικές σκέψεις. Ε, budget 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Budget 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. πέντε του προεπιλογισμού. Υπέρ. όχι. Α, συγγνώμη, συγγνώμη. Κάτι έκανα λάθος. Α, απορρίφθηκε. Τροπολογία 2 λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 3 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 4 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 5 α καταπίπτει καταπίπτει budget 6 η 6 της Επιτροπής Προπολογισμών παρακαλώ η 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και τώρα τελική ψηφοφορία όπου έχουμε διάφορες ψηφοφορίες. Καταρχάς, το σχεδίο νομοθετικής πρότασης όπως τροποποιήθηκε ηλεκτρονικά παρακαλώ, συνάδελφοι. There are two Δύο σοσιαλιστές και ένας από το ECR παρακαλώ περισσεύουν. Αφαιρέστε κάρτες. Σας παρακαλώ περισσεύουν δύο ψήφοι από τους σοσιαλιστές και μία από το ECR. Ένα σοσιαλιστής τώρα. Α, όχι. Από το ECR. Παρακαλώ, ο επιπλέον βουλευτής να αφαιρέσει την κάρτα του. Μάλιστα. Ωραία. Έναρξη ψηφοφορίας λοιπόν. Πέρας ψηφοφορίας. 37 υπέρ, 3 κατά, 5 αποχές. Τώρα το νομοθετικό ψήφισμα. Το νομοθετικό ψήφισμα ψηφίζουμε. Ηλεκτρονικά και πάλι. The vote is closed. And... Πέρας. 36 υπέρ, 3 κατά, 6 αποχές και τώρα χρειαζόμαστε απόλυτη ε, πλειοψηφία για την εντολή, για τις διαθεσμικές διαπραγματεύσεις. Μία κουβέντα επιτρέψτε μου ακόμα ψηφίζουμε για την εντολή για τις διαπραγματεύσεις, ε, η τροποποιημένη πρόταση και για την ομάδα διαπραγματεύσεων που θα αποτελείται από όλους τους κοιόδης, τον εισηγητή και την πρόεδρο της Επιτροπής. Αυτό λοιπόν χρειαζόμαστε 26 ψήφους υπέρ. Έναρξη παρακαλώ της ψηφοφορίας. The vote We have 40 people in favor, υπέρ, 3 κατά, 3 αποχές. Άρα θα ξεκινήσουν οι πραγματεύσεις. Και μετά θα περάσουμε στην Ολομέλεια. Α, όχι. Θα περάσουμε στην Ολομέλεια. Α, όχι. Μετά θα πάμε στην Ολομέλεια. Thank you. Now we go to Georgia και τώρα περνάμε στην ε, γνωμοδότηση του Γεώργιου Σταυρακάκη για τον Γενικό Προϋπολογισμό. Πολύ σύντομη θα είναι η ψηφοφορία. Τραπολογία 1 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τραπολογία 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε το σύνολο της γνωμοδότησης όπως τροποποιήθηκε. Ηλεκτρονικά παρακαλώ η ψηφοφορία. Πέρας. Σαν τέσσερις ψήφοι υπέρ, τρεις αποχές. Εγκρίνεται. Στο επόμενο θέμα, στην ημερήσια διάταξη, γνωμοδότηση Τάμας Ντόιτς για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Να ξεκινήσουμε παρακαλώ. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ, 3 λέω υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 4 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 5 αποσύρεται. 6 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 4, 5, συγγνώμη 7 υπέρ, κατά αποχές να ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά την τροπολογία 7. Έναρξη πληροφορία.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 κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα τελική ψηφοφορία παρακαλώ ηλεκτρονικά έναξη της ψηφοφορίας. Πέρασε. 43 ψήφοι υπέρ, 3 κατά, μία αποχή, συγχαρητήρια. Και τώρα περνάμε στην έκθεση γνωμοδότηση χώζα συμπράσα, σχέδιο δράση για την ηλεκτρονική υγεία. Να ξεκινήσουμε. Τροπολογία 1. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 4 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ. Να ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά την 5. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρασε. Εγκρίνεται 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ Κατά. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά στην ελέγξουμε και αυτή παρακαλώ την 7. Έναρξη ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται 22 υπέρ, 24 κατά, 8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές έγκρινεται 13 υπέρ, κατά αποχές έγκρινεται 12 υπέρ, κατά αποχές έγκρινεται 14 υπέρ, κατά, α, συγγνώμη, Για την 14 έχουμε προφορική τροπολογία. Είναι κάτι, κανείς κατά της προφορικής τροπολογίας. Όχι, όπως τροποποιείται. 14 λοιπόν υπέρ. Κατά αποχές έγκρινεται 15 υπέρ. Κατά αποχές έγκρινεται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 Εγκρίνεται 29 υπέρ, 18 κατά. Τελική ψηφοφορία, παρακαλώ ηλεκτρονικά. Έναρξη ψηφοφορία. The vote is closed. 44 ψήφοι υπέρ, μία κατά, μία αποχή. Σχεδόν ομόφωνα. Συγχαρητήρια. Και τώρα περνάμε στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο την περίοδο 2014-2020. Ανδρέη Κοβάτσεκ, στο 15, μία μόνο ψήφος. Ηλεκτρονικά, παρακαλώ, η ψηφοφορία, έναρξη της ψηφοφορίας για την ε, έκθεση Ανδρέη Κοβάτσεκ. Πέρας. 43 υπέρ, 3 κατά, μία αποχή. Εγκρίνεται συγχαρητήρια και τώρα νομίζω ολοκληρώσαμε τις ψηφοφορίες. Και εσείς, και εσείς τελειώσατε. Περνάμε λοιπόν στο 16, μιας και έχουμε εδώ όλους τους συναδέλφους, έχουμε το σχέδιο γραμματότησης ε, για την... συναδελφή στο 16 που έχουμε στην ημερήσια διάταξη. Στις 11 είπατε ότι θα ξεκινούσαμε, αλλά μιας και είναι όλοι εδώ παρόντες, νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε πάρα αυτά με το 14, με το 16, συγγνώμη. Όλτριχ, να παρουσιάσει την ομοδότησή σου. Κυρίες και κύριοι. Θα σας παρακαλέσω να φορέσετε τα ακουστικά σας. για να κάνω κάποια σχόλια για την έκθεσή μου. Αυτές οι αυτά τα σήματα περιφερειακά, σήματα ποιότητας ε, είναι αποδεκτά, ε, μπορεί να είναι γεωργικά ή μη γεωργικά, πρόκειται για σήματα τα οποία υπάρχουν παράλληλα με τα λοιπά σήματα έχουν πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ε, ταύτιση με την περιοχή και διασύνδεση. Έχουν βέβαια να αντιμετωπίσουν αρκετά σημαντικούς ε, κινδύνους και προκλήσεις. Προσθέμενη αξία. Η προσθέμενη αξία τους μπορεί να είναι η ενίσχυση του ενδιαφέροντος της ε, υπηρεσίες ή του στέγη που προσφέρεται σε μια περιφέρεια, στον τρόπο διατροφής της, στον τρόπο ζωής της και βέβαια μπορεί να έχουν από την άλλη ενίσχυσή τους ε, μπορεί να έχει συνέπειες και για το περιβάλλον ακόμα για τις συνθήκες παραγωγής. Εγώ στην εκθεσή μου επισημαίνω ορισμένε ε, παρατηρήσεις που θα παρακαλέσω να λάβει την υπόψη ε, η Επιτροπή ότι καταρχάς εφόσον υπάρχουν κίνητρα πρέπει να ομολογηθεί ότι αυτά συνεπάγονται σημαντικό γραφειοκρατικό φόρτο. Δεύτερον, ότι πολύ λίγη σημασία δίνεται στα περιφερειακά σήματα ποινότητα και ιδιαίτερα στην υποστήριξή του ε, για την ε, ένταξη στην αγορά. Πολύ λίγε είναι περιφερειακέ ή τοπικέ στρατηγικέ για την ανάπτυξή του και τη βελτίωσή του. Ε, πράγμα το οποίο θα σήμαινε βέβαια υποστήριξη από την Ευρώπη. Οργανωτικά, οι οργανώσεις οι οποίες εκπροσωπούν αυτά τα περιφερειακά σήματα ποιότητας και που τα προωθούν, οργανώσεις οι οποίες ίσως να μην περιορίζεται μόνο στην παραγωγή γεωργικών προϊόντων, είναι οργανώσεις οι οποίες δεν έχουν πάντα το απαραίτητο προσωπικό, ούτε τις κατάλληλες οργανωτικές δομές. Και επιπλέον χρειάζεται μια αποτελεσματική, μια ουσιαστική ανταλλαγή ιδεών και εμπειρίας σε επίπεδο και εθνικό και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλή ιδέα θα ήταν λοιπόν αυτές τις οργανώσεις να τις λαμβάνουμε υπόψη για τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Αυτά είχα να σημειώσω. ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Ρώσα. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και συμφωνώ με τον κύριο Βλαζάκ οποίος θέλει να υποστηρίξει την τοπική αυτή παραγωγή περιφερειακών σημάτων ποιότητας. Είναι σημαντικό βέβαια να στηρίξουμε τις προσπάθειες των επαγγελματιών. Στην έκθεσή μας όμως νομίζω δεν γίνεται λόγος για ένα νέο σύστημα ε, σημάτων ποιότητα, περιφερειακών σημάτων ποιότητα. Γιατί στη τελευταία ανάλυση η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στη θέση τη ήδη αυτές τις, ε, αυτά τα μέσα δεν χρειάζεται να εισαγιαχθεί ένα νέο νομοθέτημα, ένα νέο μέσο το οποίο μόνο θα μπορούσε να επιδεινώσει τη, συνοχή, τη σύγχυση και τα προβλήματα ως προς την αναγνωρισιμότητα. Υπάρχουν λοιπόν μέσα, μπορούμε να αξιοποιήσουμε για να βελτιώσουμε και να προαγάγουμε την ευρωπαϊκή ποιότητα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να επικεντρωθούμε στην παραγωγή ποιότητας, να προσφέρουμε κάθε δυνατή βοήθεια φυσικά και υποστήριξη από τα διαρθρωτικά ταμεία, αφήνοντας και ένα περιθώριο βέβαια για την ε, διάθεση στην αγορά και την παραγωγή σε επίπεδο τόσο ευρωπαϊκό όσο και διεθνέ εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε να προσφέρουμε λοιπόν χάρη στο ευρωπαϊκό, στην ευρωπαϊκή υποστήριξη μια προσθέμενη αξία. Ε, μιλισμονούμε ότι τα προϊόντα μας είναι προϊόντα τα οποία έχουν υποβληθεί στις πιο απαιτητικέ παληθεύσεις και δοκιμές ως προς την φυτογενή κυρίως διάσταση και γενικά επαλήθευση για τη δημόσια υγεία. Άρα και μόνο αυτή τη διάσταση να κοιτάξουμε έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Ταυτόχρονα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι από ό,τι φαίνεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τις αρχές του 2014 θα επαβάλει έκθεση για την εισαγωγή μια ειδική ονομασία ε, προελεύσεω για τι νησιωτικέ περιοχέ, Πράγμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό για τα νησιά και μπορεί να τους προσφέρει ακόμη περισσότερη υποστήριξη. Όλα αυτά τα νησιά τα οποία εξαρτώνται τόσο πολύ από τον τουρισμό και από τα τοπικά τους προϊόντα. Κάποιος άλλος ομιλητής παρακαλώ. Εκ μέρου του Σιχελιστών, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, έχεις ε, αναλάβει να αντικαταστήσει την Φραντσέσκα. Ναι, ε, η Φραντσέσκα και την αντικαθιστώ. Στη συνεργασία της με τον εισηγητή, ιδιαίτερα η Φρανσέσκα επέμεινε στην περιφερειακή διάσταση. Διάσταση η οποία θα επιτρέπει την διάκριση μεταξύ των διαφορών προϊόντων και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους. Ιδιαίτερα δε, σε ένα δεύτερο σημείο, επιμένει και στην έννοια της, ε, ε, του περιφερειακού σήματος ποιότητας, στον ορισμό, στο τι θα περιλαμβάνει αυτό, γιατί είναι αρκετά ασαφής η έννοια αυτή και η σκιώδη συγκητριά μας πιστεύει ότι θα πρέπει ε, η ενδεχόμενη δημιουργία αυτών των σημάτων, περιφερειακών σημάτων ποιότητας, δεν θα πρέπει να επικαλύψει τις ε, παραδοσιακές ε, ονομασίες προελεύσεως και ποιότητας, τα DOP, COP και το καθεξής, τα οποία έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητά τους όλα αυτά τα χρόνια. Και επίσης, για τον κύριο Βλάσακ, αυτή η προσέγγιση στο περιφερειακό σήμα πρέπει να παραμείνει κοινοτική, ευρωπαϊκή. Να μιλάμε για ένα πλαίσιο ευρωπαϊκό που θα ισχύει για όλες τις ε, περιφέρειες της Ευρώπης. Να μην αρχίσουμε διαφοροποίηση ανάλογα με περιοχή και περιφέρεια ή κράτος μέλος. Γιατί αυτό μέσα σε ένα ε, δεδομένο ευρωπαϊκό θα περιέπλεκε πολύ περισσότερο τα πράγματα και βέβαια θα έπλητε ασφαλώς και την ανταγωνιστικότητά του ως ευρωπαϊκό επίπεδο και σε διεθνές. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μπίρντερ, μέρος των Φιλελευθέρων. Ναι, Πρόεδρε. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση η σχετική με τα περιφερειακά σήματα τα οποία έχουν νομίζω κατά βάση ε, ιστορικό χαρακτήρα. Πράγματα τα οποία γίνονταν από παλιά και που προσπαθούμε να διαφυλάξουμε και να προαγάγουμε. Διερωτώ με λοιπόν, ο εισηγητής έχει αναλογιστεί πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε την παρουσίαση και νέων τέτοιων σημάτων από τις κοινότητες. Το μικρόφωνο της Πρόεδρου ανοιχτό και είναι δύσκολο να παρακολουθήσουμε τον μιλήτη. Ε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να Ευχαριστώ πολύ. Να ε, προστατεύσουμε την τοπική παραγωγή. Πρέπει λοιπόν να βρούμε έναν τρόπο να δώσουμε και την αναγνώριση και στην καινοτομία, στη δημιουργία ενός νέου προϊόντος. Ίσως αυτό το σήμα θα μπορούσε να ενσωματωθεί στο περιφερειακό σήμα ποιότητας και την έκθεση του κυρίου Βλάσακ και να δώσουμε κάποιες ιδέες για το πώς μπορούμε να ε, εντοπίσουμε νέες, νέα σήματα ποιότητας, νέα δημιουργία στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Αλφονσί. Πράσινη. Ε, πρόεδρε, ευχαριστώ. Πάντοτε υποστήριζε η ομάδα μας ε, και τη γεωργία ασφαλώ και την περιφερειακή ανάπτυξη. Τα καλύπτει αυτά η έκθεση του κύριου Βλάσσα και εμείς θέλουμε μια γεωργία που θα είναι πιο οικολογική και περιφερειακή ανάπτυξη που θα επιτρέπει και στα παραδοσιακά προϊόντα να αναδεικνύονται περισσότερο και να προστατεύονται. Λοιπόν, είμαστε υπέρ αυτών των προσπαθειών και γι' αυτό υποστηρίζουμε και τις θέσεις και την έκθεση του κυρίου Βλάσσα και είναι πλήρης πιστεύουμε. Ευχαριστώ, Μάκιν Άντερσον. Από την ΚΟΕ είναι κανείς εδώ. Κανείς από την ΚΟΕ. Και εμείς υποστηρίζουμε τις αρχές που εκθέτει η έκθεση αυτή. Όπως είπε και ο συνάδελφος Αλφόνση, γιατί πρόκειται για βελτίωση των δραστηριοτήτων. Στην Ήπεθρο τέλο πάντων υποστηρίζουμε πλήρως τους στόχους τη έκθεση. Μάλιστα. Υπάρχουν άλλα σχόλια. Η γνωμοδότηση θα ψηφιστεί στη συνεδρία μας στις 14 Οκτωβρίου, γι' αυτό έχουμε πολύ μικρή διορία για την κατάθεση τροπολογιών αλλά πληροφορήσαμε τους κοιόδης για να το κοιτάξουν. Αύριο 25 Σεπτεμβρίου στις 12 λίγη. Θέλεις να προσθέσεις τίποτε όλτσι. Μόνο να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τη συζήτηση και αν θέλουν να μου στείλουν σχόλια ευχαριστώ Ωραία πάει και αυτό. Πού είναι ο Λαμπέρ. Το 17 τώρα. Το 17 έκθεση Βανής Τελρόη και λοιπά για τις διαπραγματεύσεις η Κωνσταντς. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε. Εκπλήσωμε και ο Λαμπέρ επίσης γιατί ετοιμάζουμε τον τριμερή διάλογο, ετοιμάζαμε και ξεχάσαμε ότι έχουμε συνεδρίαση και της Επιτροπής, αλλά πάντων. Τελικά ετοιμαστήκαμε. Λοιπόν, είναι νομίζω η πρώτη μας συνεδρίαση μετά τας διακοπάς, αλλά ήδη έγιναν από τότε έξι τριμερείς διάλογοι. Γι' αυτό χρειάστηκε να ξανακάνω restart το μυαλό μου για να το καταλάβω. Λοιπόν, συζητούνται πολλά από την αιτιολογική διέκθεση και στις τεχνικές συναντήσεις υπήρξε λίγο πολύ συμφωνία με τα περισσότερα δημοσιονομικά θέματα και θα μπορούσαμε να καταλήξουμε εκτός από το αποθεματικό γιατί όπως ξέρετε From the Fishery Committee. η Επιτροπή Αλληλείας μας έστειλε μερικά καινούργια, μερικές καινούργιες πληροφορίες και δεν μπορέσαμε να τις συζητήσουμε πλήρως για να συμπεριληφθούν γιατί υπήρχαν δυσκολίες. Είδα όμως τι προτάσεις θα συζητηθούν σήμερα στον τριμερή διάλογο και θα συνεννοηθούμε. There is a rest still open in the financial instrument για τα δημοσιονομικά εργαλεία και τους εξάντε όρους. Πάλι για το σημερινό τριμερή διάλογο, αλλά σήμερα θα λήξουν αυτά, θα τα κλείσουμε. Υπάρχει ένα ευρύτερο θέμα όμως που αφορά την πρωτοβουλία για τις ΜΜΕ της Κομισιόν την περασμένη εβδομάδα αρχίσαμε να το συζητάμε. Και νομίζουμε ότι ξαφνικά η Επιτροπή ευνηδιαστικά μας έκανε μια καινούργια πρόταση και γι' αυτό και εμείς είπαμε εντάξει, αλλά αν προλάβουμε μέχρι τη δεύτερη σύνοδο του Οκτωβρίου, όπου θα ψηφιστούν όλα αυτά, αν βρούμε χρόνο να το λύσουμε, θα το λύσουμε. Αλλά αυτό θα είναι το τελευταίο σημείο, είπαμε, στις διαπραγματεύσεις. Γιατί θα μπορούσε να λυθεί αργότερα. Δεν, δεν θέτει ιδιαίτερε δυσκολίες για τις ΜΜΕ και γι' αυτό είπαμε πρώτα τα υπόλοιπα και μετά αυτό. Έχετε τα έγγραφα με ό,τι αποφασίσαμε. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αρχίσαμε να το συζητούμε την περασμένη εβδομάδα στον πολιτικό τριμερή διάλογο και φάνηκε ότι τέσσερα είναι μάλλον τα κυριότερα προβλήματα. Η performance reserve που λέμε, όπου η Κομισιόν προτείνει 5% ενώ υπήρχε πρόταση και για 7% δηλαδή 30 δισεκατομμύρια νωρίτερα να δοθούν στις περιφέρειες. Άρα πρόκειται για αναβολή για την επόμενη δημοσιονομική περίοδο μετά το 20. Μετά υπάρχει το θέμα των όρων για, την μακροοικονομη... για τις μακροοικονομικές ρήτρες και προσπαθήσαμε όλα αυτά να τα συνδυάσουμε σε μία δέσμη αλλά η μακροοικονομική όρη και η performance reserve είναι πολύ δύσκολο να συνδυαστούν και να λυθούν. Γι' αυτό θα το συζητήσουμε σήμερα για να δούμε αν υπάρχει καμία δυνατότητα να τα συνδυάσουμε και να κάνουμε ένα συμβιβασμό. Γιατί ο Μάρτιν Σούλτ και η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισαν να μην ψηφίσουμε για το Πολδίπ όσο αν δεν έχουν εγκριθεί και δια, τύχη διαπραγμάτευση ή συνθήκες ανατομέα. Αν βρεθεί κάποια συμβιβασμός για τα τέσσερα προβλήματα, καλά, αλλιώς επειδή είναι μεγάλη η πίεση, και πρέπει να βρούμε κάποιο συμβιβασμό. Δεν σημαίνει αυτό ότι οι πολιτικές μας ιδέες με πολύ μεγάλη πλειοψηφία μέχρι τώρα μπορούν να χαθούν τελείως. Πρέπει να σας πω ότι δυστυχώς η γερμανική κυβέρνηση ιδιαίτερα είναι υπέρ της μακροοικονομικών όρων αλλά δεν ξέρω πότε θα σχηματιστεί η κυβέρνηση γιατί αργεί. Γι' αυτό είναι δύσκολο το πράγμα. Άρα θα επανέλθουμε αργότερα. Ευχαριστούμε πολύ ο Λαμπέρ. Ευχαριστώ Κωνσταντ για αυτή σου την πληροφόρηση. Είχαμε πολλές συνομιλίες με την Κομισιόν και το Συμβούλιο, όλα υπόθηκαν. Μετά από 65 τριμερή διαλόγους, τι να προσθέσουμε, αυτό πρέπει να αποφασίσουμε. Πώς να συνδυαστούν όλα αυτά σε μια συμβιβαστική πρόταση. Και η διαπραγματευτική ομάδα επίσης δεν θέλει να παραμείνουν όλα σαφή και φλού και να μην καταλήγουν. Εμείς επιμένουμε κυρίως περί του Πολυδίπ. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τιμήσουμε την διαπραγματευτική μας εντολή τα σκεφτόμαστε και θα τα ξαναπούμε σήμερα στη διαπραγματευτική ομάδα. Ένα άλλο σχόλιο, κάτι που έχει ήδη γίνει για μας, έχει λυθεί, είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Από ό,τι γνωρίζω, η Επιτροπή Απασχόλησης συμμετείχε στη διαπραγμάτευση αλλά και τα είχε δεχτεί όλα αλλά σήμερα τα αλλάζει. Τα αλλάζει. Εμείς θα επιμείνουμε στο συμβιβασμό που είχαμε πετύχει για το σύνολο. Αυτό είναι το σημαντικό, να τα δούμε όλα μαζί, όχι μόνο τα ποσοστά αλλά και τους μηχανισμούς τους για το συνδυασμένη χρηματοδότηση κοινωνικού και περιφερειακού ταμείου. Αυτό δίνει πολύ μεγάλες δυνατότητες για κοινή προσέγγιση μεταξύ πόλεων και υπαίθρου. Και χθες ακούσαμε ότι υπάρχουν θετικά παραδείγματα εμπειριών. Παραδείγματος χάρη πήγαμε στο Βερολίνο πριν από τρεις εβδομάδες και είδαμε εκεί ότι η κοινή χρήση της πολυχρηματοδότησης λειτουργεί και δίνει μεγάλες δυνατότητες γιατί οι κοινωνικοί στόχοι δεν αποκλείονται από το περιφερειακό ταμείο αλλά προστίθενται σε αυτού. Όταν θα γίνει αυτή η συζήτηση τότε θα έχουμε και εμείς μια σαφέστερη θέση. Εμείς δεν πρόκειται να εμποδίσουμε καμιά διαδικασία, ούτε να σταματήσουμε τις εργασίες μας. Φαίνεται ότι στην Επιτροπή Απασχόλησης δεν υπήρξε ακόμη τελική ψηφοφορία για το Κοινωνικό Ταμείο, αλλά θα σας τα λέμε, θα σας πληροφορούμε συνοπτικά και περιληπτικά για να μπορούν οι ομάδες να τα συζητήσουν. Δεν ισχύει ότι μόνο το 25% μας ενδιαφέρει. Πολύ ευρύτερα ενδιαφέροντα έχουμε από αυτήν την άκαμπτη προσέγγιση. Αυτά σας τα λέω εν πάση ειλικρινία, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να προσθέσω δύο σχόλια για δύο θέματα. Καταρχάς, σε δύο φορά το κοινωνικό ταμείο, θα ήθελα να σημειώσω ότι πολλοί, πολλοί συνάδελφοι από τις άλλες επιτροπές παρουσιάζουν ε, τις απόψεις τους κατά τη συμφωνία που πέτυχε η διαπραγματευτική μα ομάδα. Να ξεκαθαρίσω ότι για τι ε, διαπραγματεύσει για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είχαμε καλέσει και τον πρόεδρο τη Επιτροπή ε, Απασχόληση και τον σχετικό εισηγητή. Σε όλες τις διαπραγματεύσεις λοιπόν είχαμε έναν συνάδελφο που ήταν ο Σκιώδης από την Επιτροπή Απασχόλησης για το Γενικό Κανονισμό και βρήκαμε μία συμφωνία την οποία υποστήριξε. Υποστήριξαν όλοι όσοι ανέφερα που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις ενεργά. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη η δικασία έβρεσης του συμβιβασμού και να θυμόμαστε ότι σε αυτό το επίπεδο αν ε, διοικωθεί άλλο το ταμείο θα είναι εις βάρος άλλων ταμείων. Αυτό το επίπεδο σημαίνει ότι το ποσοστό του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στο σύνολο των ε, εκχωρήσεων μιλάμε για το 1 τρίτο σε ό,τι αφορά και να θυμόμαστε ότι πρόκειται για ένα ελάχιστο όριο. Αυτό είναι πάρα πολύ σαφές ε, και περιλαμβάνεται ως όρος ε, ότι δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από το τρέχον επίπεδο. Μετά μπορούμε να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Κάποια κρατημέλη θα φτάσουν και στο 50%. Να το έχουμε λοιπόν αυτό υπόψη. Αν παρουσιαστεί ως τροπολογία στην Ολομέλεια μπορεί να μπλοκάρει όλη την ε, συμβαστική συμφωνία και θα διακινδυνεύσουμε όλη την, θα διακυβεύσουμε όλη την διαδικασία. Και το έργο φυσικά που έχει δαπανίσει και η Επιτροπή μας, γιατί αυτό που μετράει τώρα για τον κόσμο είναι από 1η Ιανουαρίου να υπάρχει ένα πλαίσιο για την πολιτική προκειμένου να μπορέσει να συνεχίσει και ο κόσμος την εφαρμογή. Άρα, να το θυμόμαστε αυτό. Δεν είναι αυτά απλά χρήματα που προέρχονται από κάπου. Όχι. Όχι. Και μιλάμε για ένα ελάχιστο ποσοστό. Συμφώνησαν δε οι πρόσωποι της Επιτροπής Απασχόλησης. Και επίσης πάρα πολύ δύσκολη η εξέφραση συμφωνία συμβιβαστική με το Συμβούλιο. Άρα θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ κακό σήμα και μήνυμα. Με όλες τις συνέπειες και δεύτερη πληροφορία. Θα θυμάστε ότι εξ αρχής αυτό Αφέ και από αυτά που είπε ο εισηγητής στην αρχή θέλαμε να πετύχουμε να γίνει ψηφοφορία στην Ολομέλεια στη δεύτερη σύνοδο του Οκτωβρίου έγιναν διαπραγματεύσει τον Ιούλιο του περσινού και θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει πλήρη συμφωνία και να έχει γίνει ψηφοφορία στις 14 Οκτωβρίου στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Αυτό θα πρέπει να γίνει λοιπόν. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει στις 10-11 το αργότερο Οκτωβρίου να έχουμε ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις. Είναι πολύ περιορισμένο το χρονοδιάγραμμα, αλλά νομίζω ότι όλοι στην ομάδα διαπραγμάτευσης και στον, ε, την, στην ομάδα τριμερού διαλόγου έχουν δεσμευτεί πραγματικά να ακολουθήσουν και να ε, αυτό το χρονοδιάγραμμα. Και επίσης αυτό που είπε η Κωνσταντσε σε ό,τι αφορά την ομάδα επαφής, ε, όπου αναφέρθηκε ότι αν δεν τα καταφέρουμε θα τα μας τα πάρουν τα θέματα αυτά σε ό,τι αφορά την μακροοικονομική αιρεσιμότητα κυρίως. Άρα είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό. Δεν μπορούμε να το διακινδυνεύσουμε, να μην υπάρξει συμφωνία. Αυτά λοιπόν από πλευράς μου, Ιβαν Σκοτμάνης. Αν μου επιτρέπετε. Να συμμεριστώ και εγώ τη σκέψη μου ως μέλος της ομάδας διαπραγμάτευσης και σκιώδης συγητής για τα δύο αυτά θέματα η μακροοικονομική αιρεσιμότητα είναι μία, ένας όρος τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το χρησιμοποιεί σαν να μας δείχνει πώς πρέπει να είναι μια χώρα για να είναι εύρωστη οικονομικά. Ωστόσο, ε, μια και ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες, η μακροοικονομική αιρεσιμότητα όπως έχει συμφωνηθεί σε ένα κείμενο απόλυτα απαράδεκτο για το Κοινοβούλιο και γιατί, διότι χαρακτηρίζει μία κατάσταση σε μία χώρα που δεν έχει μακροοικονομική αιρεσιμότητα και υπό ποιου όρου δεν θα έχει τη μακροοικονομική αιρεσιμότητα. Και λέει το εξή η πρόταση επιτροπή. Όταν μία χώρα δεν τηρεί το πρόγραμμα για τον περιορισμό του περιβολικού ελλείμματος, όπως το έχει ορίσει από την πρώτη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 50% των κονδυλίων για τη χώρα αυτή πάνε στο δοθηματικό. Δεν καταβάλλονται. Δεν εκταμιεύονται. Την πρώτη φορά που διαπιστώνεται αυτό. Τη δεύτερη φορά που διαπιστώνεται η μητήρηση του προγράμματο, ολόκληρο το ποσό πάει στο Παθηματικό. Τώρα πείτε μου, το 2011 που είχαμε 17 χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση σε κατάσταση υπερβολικού ελλείμματο, συμπεριλαμβανομένων και των μεγάλων χωρών, των πλούσιων χωρών χορηγών, και οι οποίε δεν έφτασαν στο επίπεδο του 3% ελλείμματο μέσα στα 1-2 χρόνια προβλεπόταν τι έπρεπε να έχει γίνει. Δηλαδή μιλάμε για χώρε όχι που έχουν κρίση, αλλά που έχουν ξεπεράσει το έλλειμμα. Δεν ξέρω πώ συμφωνήθηκε αυτό στο Συμβούλιο, πώ πέρασε από το Συμβούλιο αυτό. Μπορεί οι Γερμανοί να έχουν κάποιο μαγικό ραβδί ή φίλτρο. Γιατί ακόμα και οι Ολλανδοί κάτω από αυτή τη στα σπάθη βρίσκονται. Πώς λοιπόν δεν μπορούν να μας απαντήσουν, γιατί θα πρέπει να μας πει ο Επίτροπος, όταν κόβονται τα διορθωτικά ταμεία, έχουμε από την άλλη πλευρά τις δαπάνες, δηλαδή έχουμε τις δαπάνες από τη Νέα μεριά και τα διαφορετικά ταμεία. Εάν τα κόψουμε και τα δύο δεν μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση. Θέλετε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θέλει με δύο ε, βούρδουλες τα λεφτά της γεωργίας και τη συνοχή να περιορίσει τα προβλήματα. Τη γεωργία δεν μπορεί να την κόψει γιατί είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Τη συνοχή όμως τη χρησιμοποίησα βούρδουλα. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να πούμε για το αποθεματικό αυτό από επιδόσεων στην οικονομία ότι δεν συμφωνούμε και συμφωνούμε με την Κωνσταντζή ότι το μόνο που φαίνεται να έχει νόημα στην υπόθεση αυτή στο αποθεματικό δηλαδή, σε περίπτωση μετήρηση των προγραμματών λιτότητα, είναι να περάσουν τα λεφτά στον επόμενο προπολογισμό. Αυτό είναι όλο. Το 7% βέβαια μπορεί να κατανέμεται σε προτεραιότητες και αν μέχρι το 2019, ε, μέσα σε ένα χρόνο, ε, ένα χρόνο μόλις από το 2020, ορίζουν, βλέπουν τα, τα χαρτιά για το κάθε κράτος και αποφασίζουν και ορίζουν ότι δεν έχει κατηρήσει τις κατευθυντήριες γραμμές, τα ορόσημα, τα, τις παραμέτρους, ό,τι έχει οριστεί και τότε παίρνουν το 7% από τις προτεραιότητες, αλλά επιτρέπουν στη χώρα ή η περιφέρεια εν λόγω να ανακαταμνήμει με τις δικές της προτεραιότητες. Μέχρι όμως καταρτιστεί το νέο πρόγραμμα, μέχρι ότου γίνει όλη η νέα αυτή η αναδιανομή, τα λεφτά αυτά πάνε ίσως σε κάποιους δικαίωχους του εθνικού προϋπολογισμού για την περίοδο μέχρι το 20. Αλλά τα πέντε λεφτά της Επιτροπής θα γυρίσουν τα κράτη-μέλη μόνο μετά το 2020. Είναι ένας πολύ απλός μηχανισμός για το πώς μπορούν να σωθούν λεφτά από την περίοδο αυτή και να μετακυληθούν στην προσεχή δημοσιονομική περίοδο. Άλλος ένας λόγος για τον οποίο είμαστε κατά της πρότασης. Μπορεί να αποτελέσει πάντως ω ε, για διάφορε αντιπροσωπείες, γιατί βέβαια θα του πούνε άπω είναι δυνατόν να μην είστε υπέρ τη μακροοικονομική αιρεσιμότητα, θέλετε να ρίχνετε λεφτά σε ένα, άδειο σε ένα τρίπιο πηγάδι χωρί πάτο και να φεύγουν και να μην τα ξαναβρίσκετε». Ε, όχι, όμω αυτό δεν είναι επιχείρημα. Καλώς λέει ο πρόεδρος, ο κύριος Ομερσή. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Ως μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας θα ήθελα και εγώ να κάνω μερικά σχόλια. Όλοι γνωρίζουμε, έχουμε συνέστηση του ότι ο προσεχής τριμερής διάλογος, η προσεχής θα είναι σοβαρή και σημαντική και ότι μπορούμε να καταλήξουμε αν είμαστε στεναροί στις πεπιθήσεις και θέσεις μας και βέβαια και αν δεχόμαστε συμβιβασμούς. Τώρα κάτι γενικότερο. Έχουμε την εντύπωση ότι κατά κάποιον τρόπο οικοδομείται εδώ η νομολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέμα της συναπόφασης. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό πολύ σημαντικό λέγω, να είμαστε πολύ στεναροί ως προς το σεβασμό των κανόνων αυτών. Υπάρχει βέβαια πίεση χρόνου, που μας υπενθύμησε και η Πρόεδρος, αλλά είναι απαραίτητο να σεβαστούμε τις δικαιοδοσίες του Κοινοβουλίου. Και δεν μπορούμε να τα αμφισβητήσουμε όλα επειδή οι πρωτοβουλίες του Συμβουλίου μας διαταράσσουν τις εργασίες μας. Τώρα για την μακροοικονομική αιρεσιμότητα νομίζουμε ότι εδώ πρόκειται για το σοβαρότερο πλήγμα κατά της περιφερειακής πολιτικής και των διαρθρωτικών ταμείων. Πρέπει να δούμε από πού προέρχεται το θέμα αυτό. Αυτή η αιρεσιμότητα για τα διαρθρωτικά ταμεία πρωτοακούστηκε πριν από πολύ καιρό και συγκεκριμενοποιήθηκε στο σύμφωνο Σαρκοζή Μέρκελ. Ρώτησα τον Επίτροπο Χάν στον τριμερή διάλογο για το θέμα αυτό, η απάντησή του δεν ήταν πολύ ικανοποιητική. Αλλά για τα άλλα προγράμματα δεν τίθενται τέτοιοι όροι. Και θέλουμε εμείς να δούμε και πέρα από το 20, είναι σοβαρό το θέμα και χαίρομαι ιδιαίτερα που το σύνολο της Επιτροπής μας παίρνει τέτοια στεναρή θέση και κοινή. Παρ' όλα αυτά επιμένω ότι πρέπει να προχωρήσουμε και ότι ίσως να είναι δυνατόν είτε διαδικαστικά είτε με άλλο τρόπο να γίνουν προτάσεις που θα επέτρεπαν να καταλήξουμε σε συμβιβασμό. Δεύτερο σχόλιο που σχετίζεται βέβαια με το πρώτο και με την συναπόφαση αφορά την κάλπα. Θα θυμάστε ότι στις 7-8 Φεβρουαρίου υπήρχαν μερικά σημεία στην απόφαση του Συμβουλίου που δεν σέβονταν τους ισχύοντες κανόνες συναπόφασης. Έγινε διαθεσμική διαπραγμάτευση μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου και όλα τα ακαθόδη θέματα αναβλήθηκαν για να συζητηθούν σήμερα στην προσθήκη 3 στον τριμερή διάλογο. Χαίρομαι γι' αυτό. Αλλά θέλω να προσέξουμε το εξής που το αναφέρει αυτή η προσθήκη 3 και που νομίζω επαναλαμβάνει το 51 το σημείο 51 της απόφασης ΚΑΛΠ για την Μαγιώτα. Στην απόφαση λοιπόν εκείνη λεγόταν στο σημείο 51 που σήμερα επαναλαμβάνεται και συμπεριλαμβάνεται στην προσθήκη 3 ότι για τα διαρθρωτικά ταμεία χρηματοδότηση 200 εκατομμυρίων χορηγείται στην νήσο της Μαγιώτα. Όπως ξέρετε θα χαρακτηριστεί ιδιαίτερα απομακρυσμένη περιοχή τον Ιανουάριο του 2014 η Μαγιώτα. Τι σημαίνει όμως αυτό. Δεν πρόκειται για πρόσθετη χρηματοδότηση αλλά για ενιαία χρηματοδότηση που χορηγείται στη Μαγιώτα έτσι 200 εκατομμύρια. Ρώτησα την Κομισιόν και το Συμβούλιο γιατί 200 εκατομμύρια, με ποια κριτήρια, με ποιους υπολογισμούς. Γιατί όχι 100, γιατί όχι 600. Δεν έχει κανένα νόημα. Δίνουν στη Μαγιότ λοιπόν ένα καταποκοπήν ποσό και τις αρνούνται την εφαρμογή των νενομισμένων κριτηρίων. Και μας λέει η Κομισιόν ότι η Μαγιότ δεν είναι στον κατάλογο των περιοχών Node 2. Άρα δεν μπορούν να τις εφαρμοστούν τα κριτήρια για τον Edge 2. Βλέπω όμως ότι παντού προβλέπεται από την 1η Ιανουαρίου του 2014 να μπει σε αυτό το κατάλογο η Μαγιότ. Και ότι άρα προφανώς τα κριτήρια του ΝΑΤΣ 2 θα εφαρμοστούν στη Μαγιότ. Αυτά τα λέω γιατί είναι ιδιαίτερα αρνητικό αυτό το καταποκοπήν ποσό και η μη εφαρμογή των κριτηρίων για αυτή την ιδιαίτερα απομακρυσμένη περιοχή, η οποία θα επωφελούνταν σε επίπεδο 450 εκατομμύριων από την εφαρμογή των κριτηρίων. Ίσως να έχει πρόβλημα απορρόφησης όπως μας λένε, αλλά δεν μπορούμε να αποδίδουμε προθέσεις εκ των προτέρων σε μία περιφέρεια ότι δεν θα μπορέσει να απορροφήσει. Όταν δεν μπορεί να απορροφήσει ισχύουν άλλοι κανόνες. Λοιπόν, αυτά είναι στην προσθήκη 3. Είναι θέμα συναπόφασης και ελπίζω η διαπραγματευτική μας ομάδα να καταφέρει και εδώ ένα συμβιβασμό εναντί του Συμβουλίου για να διορθωθεί η αδικία αυτή. Σας ευχαριστώ. Καμιά άλλη ερώτηση, κανένα σχόλιο. Ο Λάμπερ. Να εξετάσουμε λίγο καλύτερα τα σχόλια του κυρίου Οζή και σε ό,τι αφορά την διαπραγματευτική ομάδα. Ενδεχομένως να είναι σημαντικά. Και τα σχόλια του συναδέλφου κύριου Γκουτμάνης που αναφέρθηκε στο συνομοθετικό μας έργο. Φυσικά. Αυτό, το ότι είμαστε συνομοθέτες, σημαίνει ότι θα πρέπει να πολεμήσουμε για το καλύτερο δυνατό περιεχόμενο, αλλά σε τελική ανάλυση η συνομοθεσία μπορεί να σημαίνει και συμβιβασμό. σε κάποια φάση ενδεχομένως στην ομάδα διαπραγμάτευσης να πούμε το εξής. Όταν διαπραγματευόμαστε δύσκολα θέματα όπως η αιρεσιμότητα της αγοράς είναι βασικό. Να είναι υπεύθυνο και τελικά επικεφαλής το κοινοβούλιο. Αυτό μιλάμε. Γι' αυτό μιλάμε. Δεν μιλάμε για 90 χώρες. Μία ιδέα θα ήταν να εξετάσουμε το ρόλο του Κοινοβουλίου υπό τους όρους αυτούς. Μια σκέψη. Γιατί μιλώντας για το Ταμείο Αλληλεγγύης, για παράδειγμα, 5 εκατομμύρια εδώ, 5 εκατομμύρια εκεί, υπάρχει διαδικασία σύμφωνης γνώμης του Κοινοβουλίου. Η χρήση λοιπόν της διαδικασίας συνομοθεσίας σημαίνει ότι μπορεί το Κοινοβούλιο να έχει το περιθώριο να δώσει συγκατάθεση ή όχι σε άλλες περιπτώσεις. Μια σκέψη αναφέρω απλά. Και μετά υπάρχει και η φάση της ε, εφαρμογής που δίνει επιπλέον δύναμη στο Κοινοβούλιο. Αυτά από πλευράς μου. Άλλα σχόλια. Θα ήθελα και εγώ, λέει η Πρόεδρος, να μας απαντήσει, όχι τώρα. Δεν νομίζω ότι γίνεται να απαντήσετε τώρα, αλλά σε σχέση που αυτά είπε ο κ. Σαλμαζή, να σας πω ότι εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο κάναμε μια πρόταση σε ό,τι αφορά την εφαρμοστική πράξη για τον κανονισμό της Επιτροπής του 2003 που δημιουργεί ένα κοινό σύστημα κανόνων, μια κοινή λίστα, ένα κοινό κατάλογο περιφερειακών μονάδων στην Ευρώπη. Μια ενημέρωση των περιφερειακών αυτών μονάδων. Και σε, αυτό το, σε αυτή την εφαρμοστική πράξη που θα τεθεί σε εφαρμογή μετά από 20 μέρες ε, τη δημοσίευση της στην επίσημη κυβερνήση. ΝΑΤΣ 1, ΝΑΤΣ 2 είναι η Μαγιότ. Δεν ξέρουμε λοιπόν ακριβώς γιατί έχει επιλεχθεί αυτή η οδός σε ό,τι αφορά την κοινή κατάταξη των περιφερειακών ομάδων. Όταν μιλάμε για περιοχή ΝΑΤΣ 2, γιατί δεν μπορούμε να ζητήσουμε τους πόρους με τη διαδικασία που προβλέπετε για τις περιοχές της εξόχους απόκεντρες. Γιατί από ό,τι έχουμε καταλάβει υπάρχει αυτή η ευχαίρεια για την εκχώρηση 200 εκατομμυρίων για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Θα θέλαμε να το κατανοήσουμε λοιπόν, να το συζητήσουμε λοιπόν κατά τον τριμερή διάλογο. Αν θα θέλετε να το μεταφέρετε αυτό στους συναδέλφους σας να μας εξηγήσουν δηλαδή γιατί, είναι, γιατί υπάρχει αυτή η ιδιαίτερη αντιμετώπιση της περιοχής αυτής. Άλλα σχόλια. Είναι πολύ απροβλεπτή αυτή η Επιτροπή. Προβλέπουμε χρόνο γιατί κάποια θέματα είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα και τελικά δεν ε, εξαντλούμε. Ο Γιάννα δεν ε, είναι μια στρατηγική εξόδου για να σώσω την τιμή της Επιτροπής μας. Να κάνω μία ερώτηση στους ε, συναδέλφους συζητητές και στην Πρόεδρο. Πόσο μεγάλος είναι ο κίνδυνος. Έχουμε κάποια στοιχεία τα οποία δεν είναι επιλημένα. Μακροοικονομικά. Αυτό είναι και το πρόβλημα της ε, θέσης των κρατών μελών. Πάρα πολύ άκαμπτη και δύσκολη. Όχι μόνο στις διαπραγματεύσεις, οι Λιθουανοί και όλοι φυσικά ξέρουμε ποια είναι η άποψη των κρατών μελών. Θα δούμε τι θα γίνει και μετά τι γερμανικέ εκλογέ, βέβαια. Το θέμα επίσης του αποθεματικού απόδοσης. Αλλά και άλλους κινδύνους έχουμε σε παράλληλες επιτροπές. Γιατί υπάρχει το πρόβλημα με την ΚΑΠ, με τον ορίζοντα 2020. Υπάρχουν διάφορα στοιχεία στην απόφαση που δεν έχουν επιληθεί. Το ερώτημα λοιπόν είναι Ποια είναι η θέση μας ως Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Είμαστε το βασικό στοιχείο ή μήπως είναι οι άλλοι αυτοί που είναι ακαμπτοί. Είναι και το θέμα του οδικού χάρτη για σήμερα. Αυτό αφενός. Δεύτερο στοιχείο τώρα για την Επιτροπή μας. Θα πάμε στην Ολομέλεια χωρίς ε, επιπλέον στοιχεία. Τίποτα δηλαδή από την Επιτροπή καινούργιο και τίποτα από το Συμβούλιο. Καμία καινούργια σκέψη και από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δύο εβδομάδε δηλαδή πριν από την ψηφοφορία δεν θα έχουμε καμία καινούργια προσθήκη. Ή θα συμφωνήσουμε ότι έχει ολοκληρωθεί, είτε όχι. Είναι ρητορικό ίσω το ερώτημα. Αλλά σα ευχαριστώ. Η πρόεδρο, να ζητήσω από του συζητητέ να απαντήσουν ο κύριο Πανίστερο. Που δεν είναι σαφέ ποιο αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί φυσικά όλα είναι θέμα ερμηνεία και αντίληψη. Εγώ θεωρώ ότι καλή πρόοδο σημειώνουμε. Έχουμε μια διαδικασία με την οποία μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα βασικά μας θέματα σε ένα πακέτο. Σε ό,τι αφορά το αποτέλεσμα που θέλουμε να πετύχουμε, έχουμε καλές ελπίδες. Δεν ξέρω που έγινε τα άλλα προβλήματα στις άλλες επιτροπές και πόσο μεγάλα είναι τα θέματα αυτά. Δεν έχω απόλυτη επισκόπηση. Δεν έχω όμως την εντύπωση ότι εμείς πηγαίνουμε πίσω, ότι καθυστερούμε για οτιδήποτε τέτοιο. Το θέμα είναι ότι ποτέ κανείς δεν ξέρει κατά πόσο υπάρχουν πολιτικά μηνύματα μέσω των οποίων τα πράγματα, ξέρετε, μεταφέρονται στην Ολομέλεια. Μιλάμε για μια διαδικασία πρώτης ανάγνωσης. Το θέμα λοιπόν που μας δίνει και τη δύναμη, αν θέλετε, είναι το γεγονός ότι θέλουμε να ξεκινήσουμε πρώτα Ιανουαρίου για να ξεκινήσουμε και να εγγυηθούμε από πλευρά μας το Ταμείο. Δύσκολα μπορώ να σας πω κατά πόσον στην Αλληλεία, στη Γεωργία υπάρχουν άλλα τα θέματα. Έχουμε πρόβλημα Υπήρχε έω τώρα, ξέρετε, και η προσέγγιση ότι, α, μια και έχουμε προβλήματα εμεί στην Αλγία και στη Γεωργία, ελάτε κι εμείς, ελάτε κι εσεί να κάνουμε ένα ενιαίο μέτωπο. Όχι, εμεί επιλύουμε ό,τι μπορούμε να επιλύσουμε. Δεν θα κάνουμε ένα μεγάλο συνασπισμό για να μπλοκάρουμε και να ασκήσουμε όσο δυνατόν μεγαλύτερη πίεση γίνεται. Γιατί έτσι θα αναλάβει κάποια υψηλόβαθμη ομάδα στο Κοινοβούλιο για να πετύχει τελικά συμφωνία για το πολιτεύσιο δημοσιονομικό πλαίσιο. Αν... Δεν τα πιστεύω ότι αν δεν επιληθούν όλα τα επιμέρου στοιχεία δεν θα περάσει το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Δεν το πιστεύω αυτό. Το θέμα είναι απλά να πιστούμε ότι, και να πιστούν και οι υπόλοιποι ότι κάναμε σωστά τη δουλειά μας. Η Κωνσταντζέ για το πολιτισμό πλαίσιο και την απόφαση που το αφορά. Νομίζω ότι η απόφασή μας για κάποιο συμβασμό ως προς την μακροοικονομική αιρεσιμότητα είναι σημαντική. Διότι εάν αλλάξουμε το αποθεματικό επιδόσεων επηρεάζει ετήσιους πίνακες του προϋπολογισμού βεβαίως και η μακροοικονομική ρεσιμότητα μας παρουσιάζεται με σαφή μηνύματα από το Συμβούλιο ότι χωρίς αυτήν δεν θα δεχθεί, δεν μπορεί να δεχθεί. Δηλαδή δεν είναι γραμμή αναδίπλωσης, δεν έχουν γραμμή αναδίπλωσης αυτό ή συμβασμό. Από την άλλη ξέρετε ότι έχουμε μια ευρύτατη πλειοψηφία για να ε, διαγράψουμε όλη την έννοια της μακροοικονομικής ρεσιμότητας. Πώς μπορούμε λοιπόν να τα συγκεράσουμε αυτά. Και βέβαια ο καθένας να ζητεί διεξόδους και πιθανές λύσεις, αλλά το θέμα είναι, θα έχουμε συμβασμούς ή ακόμη και χωρίς συμβασμούς ένα μέρος του Κοινοβουλίου θα ταχθεί υπέρ, ενώ κάποιο άλλο κατά. Αυτό πρέπει με πολύ μεγάλη προσοχή να σταθμίσουμε, να διαπραγματευτούμε και έτσι να πάμε να μιλήσουμε στα κράτη-μέλη, με όποιο συμβασμό έχουμε στα χέρια μας. Αλλά είναι το πιο κρίσιμο ζήτημα. Στην ε, γεωργική πολιτική πρόβλημα ως προς τα ποσά δεν έχουμε. Δεν ε, τροποποιείται στον τομέα αυτό το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, ούτε και επηρεάζεται η ψηφοφορία για το MFF ανάλογα με τις διαπραγματεύσεις με την Επιτροπή για τη Γεωργία ή τις προοπτικές 2020, η μακροοικονομική ερεσικουμότητα δηλαδή και το αποθεματικό επιδόσεων εν τέλει θα είναι αυτά και αυτή είναι δική μας απόφαση δηλαδή που θα κρίνουν όλη την απόφαση για το πολιτές πλαίσιο. Και για να το πω ξεκάθαρα, αυτό σημαίνει και πίεση από τα κράτη-μέλη προς τους ευρωβουλευτές. Θα ασκηθεί οπωσδήποτε. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε μια λύση με τον τριμερή διάλογο. Τώρα εάν στην Αλία δεν έχουν κλείσει τα θέματα μέχρι το τέλος του έτους. Υπάρχουν κάποιες ιδέες να ξεκινήσουμε με την πολιτική συνοχής. Πιο νωρί και μετά να ακολουθήσει η Γεωργία και η Ελία. Δεν είναι ζήτημα δηλαδή να ληφθεί απόφαση τώρα. Αλλά για την Ολομέλεια ξέρετε ότι χρειάζεται μία ψηφοφορία και βεβαίως Υπάρχουν διαδικασίες που βλέπω ποτέ διαδικασίες για την υποβολή μιας τροπολογίας, όπως είπε για το Κοινωνικό Ταμείο Λάμπαρτ η Επιτροπή του, της Απασχόλησης, δεν ξέρω αν θα είναι ως Επιτροπή ολόκληρη, ως ομάδα. Ε, μπορεί κανείς να στήσει τροπολογία, η οποία όμως πάλι θα κριθεί από την πλειοψηφία και ελπίζουμε ότι δεν θα ε, περάσει καμία τροπολογία στην ε, προφορική στην Ολομέλεια. Γιατί όλα αυτά προχωρούν με πολύ Προσεκτικού συμβασμούς και όσο και αν δεν είναι ιδεώδης αυτή, και το ξέρουμε, είναι ο μόνος τρόπος να ξεφύγουμε από μια κατάσταση ώστε να μπορούν και οι βουλευτές να λένε στις αρχές του 2014 είμαστε σε θέση να διαθέσουμε στις περιφέρειες τα κονδύλια για την πολιτική συνοχή που είναι και το πάρα πολύ σημαντικό και απαραίτητο. Λόγω ακριβώς της πολύ κατάστασης που γνωρίζουν οι περιφέρειες αλλά και δεδομένου ότι έχουμε ευρωεκλογέ. Από τον Απρίλιο και μετά είμαστε σε προεκλογική εκστρατεία και δεν θέλω να δώσω επιχειρήματα στους αντιευρωπαϊστέ που θα λένε ότι να, δεν μπορούν ε, ούτε να αξιοποιήσουν οι περιφέρειες, δεν μπορούν τα λεφτά που τους δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αξιοποιήσουν. Θα ήταν πολύ κακό αυτό. Ευχαριστώ, τσίκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. την χάνει να είμαι μέλος της Επιτροπής Γεωργίας. Συμμετέχω ενεργά στις εργασίες για τη μεταρρύθμιση. Έχουν κλείσει όλα τα θέματα, δεν υπάρχουν πλέον εμπόδια και μέσα στις προσεχείς ώρες, αν όχι ημέρες, ε, θα είμαστε θέση να δημοσιεύσουμε μια ανακοίνωση ότι κλείνουν οι διαπραγματεύσεις και είναι έτοιμοι για ψηφοφορία η πολιτική για την γεωργία στο Στρασβούργο. Επομένως δεν θα έχουμε στο θέμα αυτό εμπόδια. Μπορούμε να υιοθετήσουμε ένα πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο για τη γεωργία. Χωρίς όμως και να θέλω να παρασυρώμαστε από τα κράτη-μέλη που ενδεχομένω θέλουν να δείξουν ότι δεν υπάρχει κοινή γεωργική πολιτική. Υπάρχει και είμαστε έτοιμοι για αυτήν. Καλώς λέει η κυρία Χιούμπνερ, αν επιτρέπετε να επανέλθω στο γενικό ερώτημα του Γιάννου, ότι δηλαδή βεβαίως υπάρχουν όλοι αυτοί οι κίνδυνοι που μας, στους οποίους εμπλεκόμαστε και εμείς με τη μακροοικονομική ρεσιμότητα κυρίως ε, και τώρα ανταποκρινόμαστε όχι γιατί φοβόμαστε να μας κατηγορήσει κανείς αλλά γιατί όπως και να έχει χρειάζεται μια απόφαση. Οκτώβριος είναι, Νοέμβριος είναι, απόφαση θα χρειαστεί όπως και να έχει. Και επίσης θα ήθελα να πω ότι ναι, μπορούμε να συζητούμε τα όσα έχουμε να διαπραγματευτούμε με τη δουλειά που έχουμε κάνει, η οποία δεν είναι απαραίτητα ορατή πάντα. Και πολλή ακόμα δουλειά βέβαια πρέπει να γίνει σε σχέση με τα... Ε, με τις αιτιολογικές αναφορές και δουλειά ως προς το νομοτεχνικό τμήμα που θα αναλάβουν οι νομομαθείς ε, γλωσσολόγοι, οι γλωσσομαθείς μάλλον νομικοί, ε, πολλά λοιπόν έχουμε να κάνουμε ακόμη, αλλά έχουμε προχωρήσει και έχουμε κάνει την ε, δουλειά στο βαθμό της ευελιξίας που μπορούμε να έχουμε. Στη μακροοικονομική όμως ερεσιμότητα ξέρω ότι κυκλοφορεί εν γέννη η φήμη ότι εγώ είμαι υπεύθυνη για την ε, απουσία πρόοδου. Ε, κατ' και ε, είναι και κομπλιμέντο, είναι και αυροφροσύνη μου λένε ότι εγώ μόνη μπορώ να το εμποδίσω. Όλοι, πάση περιπτώσει, όμως το, το βασικό μήνυμα που θέλω να περάσω είναι ότι χρειάζεται να προχωρήσουμε. Καλώς. Εάν δεν υπάρχουν άλλα σχόλια, μπορούμε να κλείσουμε το θέμα αυτό, που ήταν και το τελευταίο για το πρωί μας. Ελπίζω να σας δω το απόγευμα αριθμούς, με περισσότερους θα έλεγα ακόμη παρισταμένους. Έχουμε ακροάσει τα κράτη-μέλη, πολύ κόσμο που θα έρθει. Σας παρακαλώ λοιπόν να είσαστε εδώ στις